μου έχει απολεστεί. Βάλτε λοιπόν και μία ψήφο δική μου παραπάνω. Μήπως κάποιος προσπάθησε να κλέψει την ταυτότητά σας και ψηφίζει με τη δική σας κάρτα. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Άλλο ένα διαδικαστικό του κυρίου Ταβάρες. Άλλη μία κάρτα που δεν λειτουργεί. Είναι καινούργια όμως, μάλλον η συσκευή θα έχει πρόβλημα. Δοκιμάστε σε ένα άλλο μηχανάκι. Ευχαριστώ πάντω. Okay, Ελπίζω η τεχνική μου συμβουλή να διευκολύνει την ψηφοφορία σας, λέει η πρόεδρο. Θα το λάβουμε υπόψη στην τελική ψηφοφορία και θα το υπολογίσουμε αν χρειάζεται ε, να, να προσθέσουμε επιπλέον ψήφο. Επόμενη ψηφοφορία, μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Schengen ΣΥΣ 1 στο σύστημα ΣΥΣ 2. Τώρα ψηφίζουμε για την τροποποίηση της απόφασης 2008-839. Το ΕΛΚ προτείνει να ψηφίσουμε on block. Συμφωνείτε, συμφωνούν και οι άλλες ομάδες. Μία ψηφοφορία λοιπόν για όλες τις τροπολογίες. Η υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνονται οι τροπολογίες και περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay. Εψήφισαν όλοι. Τώρα λειτουργεί και η συσκευή του κ. Ταβάρες. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. 36 υπέρ, γιατί προσθέτουμε και τον κύριο Αλβάρο. Μία ψηφο, κατά, μία αποχή, μεγάλη πλειοψηφία και πάλι. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία δικτύου αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης. Ο κύριος Δίας Δεμέρα είναι ο εισηγητής. Okay. Με πληροφορούν ότι είναι ενδεικτική η ψηφοφορία μόνο, γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις και θέλουμε απλώς να γνωρίζει ο εισηγητής ε, πώς θα ήταν σκόπιμο να μας εκπροσωπεί στις διαπραγματεύσεις. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία με την τροπολογία 8 της κυρίας Κέλλερ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο εγκρίνουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Για να το επιβεβαιώσουμε, συγγνώμη. ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Όντω, απορρίπτεται. 21 ψήφοι κατά, 17 υπέρ και μία αποχή. Τροπολογία 9 ναι, έχει αποσυστεί. Τροπολογία 10 της κυρίας Κέλλερ, ψήφι υπέρ, κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. Τροπολογία 11 της κυρίας Κέλλερ. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 της κυρίας Κέλλερ. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της κυρίας Γκυγιόμ. Υπέρ, κατά, αποχές, Να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. 14 έχει αποσυρθεί, 16 ψήφοι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές και πάλι να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορία. 22 υπέρ, 18 κατά. Τροπολογία 15. στη υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. Σαφώς απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το ελέγχουμε γιατί δεν μπορούμε να δούμε αν είναι υπέρ ή κατά. Έρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 22 υπέρ, 18 κατά. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Να το ελέγξουμε. Η τροπολογία 20 ψηφίζουμε. «22 υπέρ, 18 κατά, η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται». Τροπολογία 18, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Α, συγγνώμη, 23. Πρέπει να αλλάξω τα γυαλιά μου, λέει η πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται όντως. Προσθέτουμε και την ψήφο του κυρίου Άλβαρο, αλλά απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Όχι 22, 24. 24, έχετε δίκιο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω να το ελέγξουμε. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά το ελέγξουμε. 22. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 25 έχει αποσυρθεί. 2 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Καταπίπτει. Τροπολογία 5. Είστε όλοι σε γρήγορη σήμερα το πρωί. Τροπολογία 5 υπέρ. Σηκώστε τα χέρια σας όλοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Εξήθησαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορία. 22 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, α, καταπίπτει 7. Θα κάνουμε τελική ψηφοφορία παρόλα αυτά. Είναι ενδεικτική ψηφοφορία είπαμε. Λοιπόν, για όλη την έκθεση ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται με μία ψήφο κατά. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Το σημαντικό είναι ότι συμφωνούμε. Όχι εγκρίνεται, αφού είναι ενδεικτική ψηφοφορία, αλλά συμφωνούμε. Καλή τύχη στον εισηγητή για τι διαπραγματεύσει. Η επόμενη έκθεση του κυρίου Ταβάρη για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης. Η πρόταση του εισηγητού και των σχεδόν εισηγητών είναι να κάνουμε τροπολογία on block. Και πάλι ενδεικτική ψηφοφορία. Όχι, όχι, επιβεβαιωτική ψηφοφορία. Επιβεβαιωτική ψηφοφορία, εντάξει. Έλεγε ενδεικτική. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές, μία αποχή, μία ψήφος κατά. Θα κάνουμε και μία τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Σύντομη ψήφο του κ. Άλβαρο, 39 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κ. Ταβάρες. Μην με μπερδεύετε. Καλά τα πάω, λέει η Πρόεδρος. Επόμενη έκθεση του κυρίου Ταβάρες. Κατάλογος ψηφοφορίας για την επιβεβαιωτική ψηφοφορία διαβάζω τώρα. Τέλος πάντων, δεν θα σας τα διαβάσω όλα αυτά. Τώρα πάντως ψηφίζουμε για το αποτέλεσμα της ε, ενδεικτικής ψηφοφορίας. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με δύο ψήφους κατά. Και κάνουμε τώρα την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη συνολική έκθεση. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή. Και περνάμε στη ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Γκάλ για την ε, ε, για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Τροπολογία 1 της κυρίας Βαζά Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αυτή η τροπολογία είναι κρατάει τρεις σελίδες βλέπω εδώ τροπολογία 2 με προφορική τροπολογία μπορούμε να ψηφίσουμε με τις προφορικές τροπολογίες όχι ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άλλη μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2 της κυρίας Χαουτάλα υπάρχουν αντιρρήσεις όχι ψήφι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της κυρίας Βεργιά, υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Σαφώς απορρίπτεται. Τροπολογία 4, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 με προφορική τροπολογία. Δεν έχουμε αντιρρήσεις. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Όχι, καταπίπτει. Γιατί τι είχαμε τη συμβαστική τροπολογία. Τροπολογία 8, ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να τα ελέγξουμε. Ωραία. Τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Όντως εγκρίνεται. 25 υπέρ, 18 κατά. 10 κατά πίπτη, Τροπολογία 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Καταπίπτει. 14. Καταπίπτει. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 4. Όχι. Α, την τροπολογία 18 δεν καταπίπτει. Τροπολογία 18. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Όχι, αυτή καταπίπτει και η άλλη καταπίπτει. Τροπολογία 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. 25 με την ψήφο του κ. Αλβάρα, έναντι 18 εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ. Για την 24. Αν δεν σηκώνετε το χέρι σας δεν μπορούμε να σας δούμε. ψήφι κατά. Πολύ καλά τώρα. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά το ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Όντως εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ, 18 κατά. Συμβαστική τροπολογία 5 ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29 με προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορία. 41 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Περνάμε στην έκθεση της κυρίας Παπαδοπούλου κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία on block. Όχι. Τις τρεις πρώτες. Τη 2 και 3 να τις ψηφίσουμε μαζί. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Για την παράγραφο 9 για το αρχικό κείμενο ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές. Κάποιος έχει αμφιβολίες για τον κατάλογο ψηφοφοριών της ομάδας. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 9. Λέει αρχικό κείμενο από την εισηγήτρια. Τροπολογία 9. Εψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 20 υπέρ, 17 κατά. Παράγραφος 11, αρχικό κείμενο από την εισηγήτρια. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την παράγραφο 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα ψηφίσετε κι εσείς, αγαπητή γειτόνισσα. Πέρασε της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 4 έχει αποσυρθεί. Προφορική τροπολογία στην παράγραφο 12 από το ΕΛΚ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5 της κυρίας Βίκστρομ, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 σε δύο τμήματα. Κατόπιν αίτηση των φιλελευθέρων για το πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 41 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Παπαδοπούλου. Και νομίζω ότι τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Μπράβο μας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε πιο αποτελεσματικοί από όσο νομίζαμε και εμείς οι ίδιοι. Hey, um, colleagues, that brings us to the next subject. Περνάμε στο επόμενο θέμα, αγαπητοί συνάδελφοι, που είναι σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία. Παρακαλώ τις συζητήσεις εκτός αιθούσης. Okay. Can we please take our seats and resume the debate and switch off our phones? Καθίστε, κλείστε τα τηλέφωνά σα για να ξαναρχίσουμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο 11 τη ημερησία διάταξη. σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία. Κατάργηση της απόφασης πλαίσιο 2004-68. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αντζελίλη από το ΕΛΚ. Είναι η πρώτη συζήτηση που κάνουμε για αυτό το θέμα. Είναι πρόταση τη Επιτροπή για οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση τη σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία. Και αυτή η πρόταση καταργεί την απόφαση πλαίσιο από τον ε, προηγούμενο πυλώνα που ε, καταπίπτει μετά την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας βασίζεται στα αρθρα 82-83 της συνθήκης. Είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα και πολύ ευαίσθητο θέμα. Και γι' αυτό χρειάζεται την ιδιαίτερη προσοχή της Επιτροπής Λίμπε και του Κοινοβουλίου γιατί μιλάμε για την προσέγγιση νομοθεσιών των κρατών μελών σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα. Είναι μια πρόταση με πολλές ε, προεκτάσεις. Η συγκήτρια κυρία Αλτζελίλη η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα κάνουν μια αρχική παρουσίαση του θέματος και θα δώσω το λόγο καταρχήν στην εισηγήτρια, την κυρία Αντζελίλη. Και μετά θα ζητήσω από την Επιτροπή να λάβει το λόγο και ελπίζω στα μεταξύ να έχουν έρθει και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Γιατί ψηφίσαμε τόσο γρήγορα, πήγε τόσο καλά η ψηφοφορία που ξεκινάμε και δεν έχει έρθει ακόμη το Συμβούλιο. Κυρία Αντζελίλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε παρουσιάζοντας την πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και την εκμετάλλευση των παιδιών και ανηλίκων και την παιδική πορνογραφία, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές οι ευχαριστίες δεν είναι οι τυπικές ευχαριστίες, αλλά επί της ουσίας, διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλεσε εξαιρετικό έργο και πραγματικά υπέβαλε μια καλή πρόταση. Η πρόταση αυτή θέτει ως στόχο την κατάργηση, την αντικατάσταση μάλλον της απόφασης πλαισίου του 2004 και τον σχεδιασμό μιας νέας νομοθετικής πράξης που να δίνει κάποιες συγκεκριμένες προτεραιότητες σε κάποια θέματα. Πρώτον, βελτίωση της ποινική δράσης κατά των αυτούργων των εγκληματικών ενεργειών. Δεύτερο, προτείνεται σκοπιμότερη και ε, πιο επίκαιρη προστασία των θυμάτων των εγκληματικών ενεργειών. Τρίτον, η πρόταση αυτή έχει σκοπό να προτείνει μια πιο διευρυμένη στρατηγική ως προς την πρόληψη των εγκληματικών ενεργειών και σε ό,τι αφορά τις μη νομοθετικές πτυχές. Τώρα ως προς το ποινικό πλαίσιο στόχος είναι να θεωρείται ως εγκληματική ενέργεια οποιαδήποτε σοβαρή μορφή κακοποίησης. Κάποιες που αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία μας. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Στη νέα πρόταση προβλέπεται η εγκληματική ενέργεια του grooming. Δηλαδή η παρουσίαση σε στο διαδίκτυο με στόχο την εκμετάλλευση. Εδώ υπάρχει και μια πιο επικαιροποιημένη, ένας επικαιροποιημένος ορισμός της παιδικής πορνογραφίας. Ένας ορισμός που καλύπτει και τις επιβαρυντικές συνθήκες που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση και την εκμετάλλευση των ανηλίκων ε, με σκοπό την ε, πορνογραφία. Αυτό δεν είναι κάτι που το προέβλεπε τόσο ξεκάθαρα η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, οι εγκληματικές ενέργειες για την εκμετάλλευση που σχετίζονται με το εξωτερικό, ο πορνογραφικός ε, τουρισμό, ο σεξουαλικό μάλλον τουρισμό, είναι κάτι που επίση περιλαμβάνει η νέα πρόταση. Επίση για το περιεχόμενο online, στο διαδίκτυο. Εδώ Συμμερίζομαι την πρόταση της Επιτροπής βεβαίως, αλλά στόχος είναι να, να αναλάβουμε δράση σε δύο μέτωπα. Πρώτα απ' όλα, με ιδιαίτερη ταχύτητα ώστε να εμποδίσουμε την πρόσβαση σε ιστότοπους που περιέχουν ε, πορνογραφικό υλικό και έπειτα να αποσπάσουμε την εξάλληψη των ε, σελίδων, των σελίδων από το διαδίκτυο που μπορεί να περιέχουν τέτοιο πορνογραφικό υλικό. Συνολική λοιπόν καταπολέμηση του πορνογραφικού υλικού που περιλαμβάνει παιδιά στο διαδίκτυο. Θα περιοριστώ σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση, καθότι είμαι πεπισμένη ότι θα έχουμε πολλές ε, παρατηρήσεις και ιδέες προκειμένου να συζητήσουμε. Να επαναλάβω ότι δεν έχουμε να κάνουμε μια πρόταση λεπτομερέστατη, ιδιαίτερα επικαιροποιημένη, και περιλαμβάνει και κάποιες καινοτόμες πτυχές. Νομίζω η πρόταση αυτή λαμβάνει πραγματικά ιδιαίτερη μέρημνα για το συμφέρον και το όφελος των ανηλίκων. Βεβαίως, ευχαρίστω θα ακούσω και τις προτάσεις και παρατηρήσεις των συναδέλφων και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης θα ακούσω και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αντζελίλη. Να καλέσω πρώτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Δεν έχω το όνομά σας δυστυχώς. Δεν γνωρίζω ακριβώς το όνομα του ομιλητή της Επιτροπής. Παρακαλώ συστηθείτε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είμαι ο Ρενάλ Πρίβε. Είμαι διευθυντής για την ασφάλεια καθώς και τις πολιτικές ελευθερίες και την ασφάλεια των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ζητήσω συγγνώμη από σας, Πρόεδρε, και τα μέλη της Επιτροπής σας, που ίσως καθυστερημένα ασχολούμαστε με το σημείο αυτό. Εάν θέλετε όμως, να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για την πρόταση της Επιτροπής. Παρόλο που παρατηρήσω ότι η συγκήτριά σας ήταν ιδιαίτερα θετικά διακείμενη. Ίσως όμως και εγώ καλό θα ήταν να δώσω κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την πρόταση αυτή και σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς, όταν μιλάμε για σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, εννοούμε και έχουμε υπόψη είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δηλαδή, την ανάγκη να καλύπτονται, μάλλον το να εμποδίσουμε σεξουαλικές ανάγκες ε, και να γίνονται αντικείμενο εμπορίας τα παιδιά με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τραυματικές εμπειρίες και να τους σωματεύουν ε, τέτοιες καταστάσεις για όλη τους τη ζωή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει από την προηγούμενη πρόταση για μια απόφαση πλαίσιο για το ίδιο ακριβώ θέμα, την οποία είχαμε υποβάλει τον Μάρτιο πέρσι. και η οποία θα πρέπει να, δεν θα τεθεί σε ισχύ ε, λόγω τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έχει γίνει λοιπόν παροχημένη η πρόταση αυτή, γι' αυτό και χρειάζεται και να υποβάλουμε μια ανανεωμένη πρόταση. Η πρόταση λοιπόν που έχετε μπροστά σα έχει στοιχεία και παλιότερα και νεότερα. Σε, πολλούς, σε πολλές περιπτώσεις συμφωνεί με την περσινή πρόταση αλλά σε ό,τι αφορά τα νέα της στοιχεία ακολουθεί μια πιο συνολική προσέγγιση, όπως την, ε, ε, την προσφυγή για, την, για τα εγκλήματα αυτά στη δικαιοσύνη, τις ποινές και συμπεριλαμβάνει στο υπάρχον νομικό σύστημα, τα συμπεράσματα της σύμβασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και νομίζουμε ότι προσφέρει και περισσότερη προστιθέμενη αξία. Εδώ πλέον αναλαμβάνουμε δράση σε πολλά μέτωπα. Πρώτα απ' όλα, γενικό στο ποινικό δίκαιο για σοβαρά εγκλήματα κατά των ε, παιδιών με την, σε σχέση με την σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση. Πολλά από αυτά θα γίνονται αντιληπτά ως ποινικά δικήματα πλέον, κάτι που δεν συμβαίνει ήδη. Τώρα, για το περιβάλλον των ε, τεχνολογιών ε, πληροφορίας και τεχνολογίας, όλες οι ανάλογες δράσεις που περιλαμβάνουν το διαδίκτυο μαζί με το grooming και την παρουσίαση του παιδικού πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο θα θεωρούνται εγκληματικέ ενέργειε. Επίση, θα προβλεφθεί μια σειρά από διατάξει οι οποίε θα έχουν να κάνουν με την ε, έρευνα των εγκληματικών ενεργειών και την ε, συλλογή στοιχείων σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσει τα στοιχεία του το το παιδί. Έπειτα, κανόνες που ισχύουν για τις δικαιοδοσίες θα χρησιμοποιηθούν για να διωχθούν οι αυτούργοι ακόμη και αν ε, έχουν εξάγει τα εγκληματικέ του ενέργειε σε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, σεξουαλικό τουρισμό δηλαδή. Έπειτα, νέε διατάξει ώστε για τα παιδιά να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα 11 μέσα και να μην υποφέρουν κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους. Περιορίζουμε λοιπόν λόγω χάρη τον αριθμό των συνεντεύξεων με τα παιδιά, των ανακρίσεων και τους δίνουμε και τη δυνατότητα νομικής ε, αρρωγής. Έπειτα ιδιαίτερα προγράμματα για την προστασία των παιδιών και επίσης ε, για την πρόληψη νέων εγκληματικών εργειών από τους ίδιους αυτούργους. Τέτοιε δράσει θα πρέπει να εξαλειφθούν από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θέλουμε να εμποδίσουμε την πρόσβαση σε ιστότοπου που περιλαμβάνουν ε, παιδικό πορνογραφικό υλικό και πολλέ φορέ εντράζονται εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μπορεί να χρειαστεί και παρέμβαση των αστυνομικών αρχών κάποιε φορέ. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία. Πρόεδρε, που προβλέπονται για την ανανέωση της ε, οδηγίας. Να αναφέρω και κάποια ακόμη, τα οποία τα θεωρώ σημαντικά. Ως προς την ανανομένη πρότασή μας. Στόχος είναι να έχουμε ένα σαφέστερο ορισμό της ε, παιδικής ε, πορνογραφίας, και τι σεξουαλικέ κακοποίησει και να προβλέψουμε και κάποιε ελάχιστε ποινέ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για, τις, για τα 22 εγκλήματα που προβλέπονται. Θα έχουμε πέντε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματο. Θέλουμε μια πιο διεξοδική διάταξη ώστε να προβλέπετε το τι σημαίνει παρέμβαση στη σεξουαλικότητα των εφήβων και επίσης να αντιμετωπίσουμε και την ύπαρξη σελίδων με πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Επίσης, συμπληρωματικές δράσεις ώστε να αντιμετωπιστεί και η πηγή. Ε, του πορνογραφικού υλικού. Γιατί όταν αρχικά υποβλήθηκε η πρόταση υπήρξαν πολλές παρανοήσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε την φραγή των σελίδων αυτών αντί για εξάλληψη. Είναι διαφορετικά τα δύο πράγματα αυτά. Η απαγόρευση της πρόσβασης είναι κάτι που μπορεί γενικότερα να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την παιδική πορνογραφία. Η εκμετάλλευση και η κακοποίηση λοιπόν των παιδιών σε σεξουαλικό επίπεδο είναι κάτι που απασχολεί όλους μας τους πολίτε. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αναλάβουμε δράση σε όλα τα επίπεδα. Η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν ε, καλωσορίσει την πρότασή μα και τη στηρίζουν ενεργά. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι και στο Κοινοβούλιο υπάρχει ιδιαίτερη ενδιαφέρον για την προστασία των παιδιών. Και πράγματι, όταν υποβάλαμε αρχικά την πρόταση αυτή, η Επιτροπή εμπνεύστηκε κατά το σχεδιασμό τη από τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 3 Φεβρουαρίου τη περσινή χρονιά που ανέθεσε στο Συμβούλιο να αντιμετωπίσει τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών. Το, το Κοινοβούλιο κατάρτισε έναν μακροσκελή κατάλογο για δράσει που πρέπει να αναλυθούν και αυτό τον σωματώσαμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην πρότασή μας που με, το νομικό ε, με την νομική τη φύση θα επιτρέψει να βελτιωθεί και η εθνική νομοθεσία των κατομελών. Τέλο, Πρόεδρε, μαζί με την πρόταση για την εμπορία αυτή θα είναι μια από τις πρώτες ευκαιρίε του Κοινοβουλίου να αναλάβει το ρόλο του ως συνομοθέτη. Εδώ έχουμε μια σημαντική βελτίωση προκειμένου να διασφαλίσουμε δημοκρατικό και δημόσιο διάλογο για τέτοια σημαντικά ζητήματα όπω το ποινικό δίκαιο και η εκμετάλλευση των παιδιών. Το νέο θεσμικό πλαίσιο ελπίζουμε θα μα οδηγήσει σε βελτίωση και επί τη ουσία τη νομοθεσία. Οι συμπολίτε μα περιμένουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την προστασία των ιδίων και των παιδιών τους από τα σοβαρότερα δικήματα και εγκληματικές ενέργειες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρίβε. Το Συμβούλιο. Παρακαλώ να λάβει το λόγο. Δεν έχω το όνομά σας. Δυστυχώς θα πρέπει να μας πείτε το όνομά σας. Αλλά δεν έχει έρθει εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Μπορούμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Τρεις συναδελφοί ζήτησαν το λόγο. Η κυρία Βίξτρομ πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προτίζει η Επιτροπή κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και όλοι το πιστεύουμε. Όποια και να είναι η ομάδα στην οποία ανήκουμε, το να καταπολεμήσουμε σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών είναι μία πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα για όλους. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει σύνορα. Ταξιδεύει παντού. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Ένα τέτοιου είδους διαζωνσιακό έγκλημα είναι κάτι το οποίο απαιτεί υψηλού επίπεδου συνεργασία μεταξύ Διότι σίγουρα θα συμφωνήσουν όλοι όταν λέω ότι θα είμαστε ισχυρότεροι αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Υπάρχουν στην πρόταση κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες θα πρέπει παρόλα αυτά να εξετάσουμε και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διάλογο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή μπορούν να συνεισφέρουν σε περαιτέρω βελτιώσεις του κειμένου. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με το πώ η Επιτροπή μπορεί να πει ότι δεν χρειάζεται εξωτερική πραγματομοσύνη όταν συγχρόνως λέει ότι δεν έχουν ακριβείς και επαρκείς στατιστικές. Αυτό για μένα είναι κάπως παράλογο και θα ήθελα να το σχολιάσει το θέμα αυτό η Κομισιό. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι είναι υπέρ του να μπλοκάρει ε, κανείς τις ιστοσελίδες που επιτρέπουν στο ίντερνετ την πρόσβαση πορνογραφικό υλικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε στη Σουηδία με συνεργασία με τους ε, ε, παρόχους ίντερνετ και με την αστυνομία. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αφήσει η Κομισιόν σε κάθε χρόνο. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια πιο γενική παρατήρηση. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότεροι δράστες τέτοιου εγκλημάτων ε, δεν μπορούν ε, να ευρεθούν από τις αρχές αλλά είναι πάρα πολύ κοντά πολλές φορές το παιδί. Μπορεί να είναι κάποιος από το οικογενειακό του περιβάλλον, το συγγενικό, ενήλικες, ε, ακόμη και κάποιος από το σχολικό περιβάλλον. Θα πρέπει να μπορεί κάπου να στρέφεται το παιδί για να μπορεί να ζητά προστασία. Οι σεξουαλικές χρήση στο ίντερνετ πρέπει να καταπολεμηθούν, αλλά συγχρόνως πρέπει να γίνει το ίδιο και στον περίγυρο του παιδιού, στο οικογενειακό ή συγγενικό περιβάλλον. Και εκεί ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Χαιρετίζω, συνάδελφοι, την πρόταση της Επιτροπής και της Επιτρόπου Μάλστρομ και θα ήθελα να συνεργαστώ στενά με την κυρία Αντζελίλη και με άλλους και όλους καθώς και με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να μπορέσουμε αυτό το κακούργημα που πλήττει αθώα παιδιά ανά το κόσμο να το καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπούσκοτ. Thank Αντικαθιστώ την σκιώδη συγητή την Μπέλκα Σίπελ που πηγαίνει προς τις Ηνωμένε Πολιτείες. Γι' αυτό εγώ την αντικαθιστώ. Πρώτα απ' όλα Αντίδεστο άρθρο 21 της πρότασης της Επιτροπής για να μπλοκάρουμε ή να αφαιρέσουμε τις ε, σελίδες του ίντερνετ του πορνογραφικού περιεχομένου. Εάν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει σύντομα, το ε, το μπλοκάρισμα αυτών των ιστοσελίδων θα μπορούσε για κάποια ε, μεταβατική περίοδο να χρησιμοποιηθεί. Όσον αφορά την πρόληψη, πιστεύω ότι δεν μπαίνει σε λεπτομέρειε η πρόταση Επιτροπή. Και η ερώτησή μου είναι προ την Επιτροπή, έχετε την πρόθεση, τι έχετε την πρόθεση να κάνετε για να προλάβετε τέτοιου είδου καταστάσει σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Δεν θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να υποχρεωθούν να υπογράψουν μια σύμβαση στην προστασία των παιδιών. Επίσης, από ποια ηλικία και μετά ένα παιδί συνενεί. Πριν από τα 18. Ποια είναι λοιπόν η ηλικία η σωστή. Αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 2. Όσον αφορά λοιπόν το grooming, το ψάρεμα των παιδιών μέσω ίντερνετ. Αυτό θα πρέπει να τιμωρείται. Αλλά πώς μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει τις προθέσεις κάποιου, πώς μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, το οποίο δυνητικά θα οδηγήσει σε σεξουαλική κατοποίηση. Τελευταία ερώτηση για το θέμα των standards για τα διάφορα, ε, για την ποινικοποίηση όλων αυτών των αδικημάτων. Ποια είναι κατά την Κομισιόν τα minimum standard. Είναι αυτά ε, συμβατά με την ε, νομοθεσία κάθε χώρας. Θα πρέπει να ζητήσουμε εναρμόνιση και πώς έχει σε τέτοιου είδους θέματα το κάθε εθνικό δίκαιο. Ευχαριστώ η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι με το στόχο της πρότασης. Το ερώτημα είναι πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και ποια είναι τα ε, ενδεχομένως κάποια αρνητικά αποτελέσματα της όλης απόφασής γιατί όλα πάντα δεν είναι ερώτημα. Τώρα, το να μπλοκάρουμε ή να φιλτράρουμε την ε, πρόσβαση πορνογραφικό υλικό δεν είναι η καλύτερη λύση διότι με πολύ λίγες γνώσεις και με δύο-τρία κλικ μπορεί κανείς να ξεπεράσει και τα φίλτρα και τις απαγορεύσεις. Νομίζω ότι όπως είπαν και κάποιοι με ένα κλικ το καλύτερο θα ήταν να μπορούμε να τα εξαφανίσουμε τα πάντα. Πιστεύουμε ότι ούτως ή άλλως οι ε, ιστοσελίδες πορνογραφικές είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα βρίσκεται παντού. Ούτως ή άλλως έχουμε συνεργασία με τις χώρες ε, οι οποίες ε, αφορώνται από αυτό το πρόβλημα και ξέρουν πώς να μπορέσουν να βρουν κάποια λύση. Ούτως ή άλλως το να αφαιρέσει κανείς την σχετική ιστοσελίδα και το περιεχόμενό ότι είναι πιο αποτελεσματικό, διότι το φίλτρο είναι μια προσωρινή λύση. Γιατί λοιπόν η Επιτροπή δεν εστιάζει να ενδιαφέρει του περισσότερου αυτό. Πώ λέτε, τα κράτη-μέλη, είπατε ότι γιατί λέτε ότι πρέπει να μπλοκάρουν τα... στι ισοσελίδε αυτέ παρά να προσπαθήσουν να τι διαγράψουν. Επόμενη ερώτηση. Ποιο νομίζετε ότι πρέπει να αποφασίσει ποιε είναι, είναι οι ιστοσελίδε που πρέπει να φιλτραριστούν και ποιε όχι. Διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε Ε, εάν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση, ε, ποιος είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει και με ποια ευαισθησία να μπλοκαριστούν κάποιες ιστοσελίδες. Επίσης, η ηλικία ε, συνένεσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, ξέρουμε ότι δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται ενδεχομένω οι κλινικέ σχέσει για νέου κάτω από 18. Είναι κάτι το οποίο ισχύει, αλλά και συμφωνώ με την κυρία Λίσκφορντ και που λέει ότι πολλέ φορέ υπάρχει και κίνδυνο για τα παιδιά από το καθημερινό του περιβάλλον. Για αυτό το θέμα, τι προβλέπει να κάνει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Κέλλερ. Τρει άλλοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Να είναι οι συνάδελφοι, παρακαλώ, σύντομοι. Κυρία Ρομέρο, πρώτα απ' όλα. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να επιμείνω στο σημείο το οποίο έθιξε και η προλαλήση σας, συνάδελφος. Διότι το σχόλιο της Επιτροπής για το μπλοκάρισμα ή για την διαγραφή της ιστοσελίδας δεν ήταν σαφές. Δεν ξέρω γιατί η Κομισιόν έκανε αυτό το σχόλιο για την ε, διαγραφή κάποιων ιστοσελίδων και θα ήθελα να μου πει ποια είναι η άποψή της. Γιατί δηλαδή δεν μπορούν να διαγραφούν αυτές οι σελίδες. Δεύτερον, που νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω. Τα δεδομένα. Σίγουρα δεν έχουμε δεδομένα για την πορνογραφία, αλλά δεδομένου ότι προσπαθούμε να συστήσουμε ένα παρατηρητήριο για την κακοποίηση και κακομεταχείριση των γυναικών, θα μπορούσαμε σε αυτό το παρατηρητήριο να συμπεριλάβουμε και αναζήτηση δεδομένων για να ξέρουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον πόσο δεδομένο είναι αυτό το φαινόμενο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στατιστικές. Γιατί αν δεν έχουμε στατιστικές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και το να έχουμε συγκρίσιμες ε, στατιστικές θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα, το θέμα της ε, ε, καταγγελίας είναι επίσης σημαντικό. Τα παιδιά δύσκολα μπορούν να καταγγείλουν μία τέτοια κατάσταση. Και είπαμε ότι πολλές φορές στο οικογενειακό τους περιβάλλον συμβαίνει ένα τέτοιο φαινόμενο. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες ε, αρχές ε, οι οποίες να εγγυώνται ε, κάποια πράγματα για να γίνεται η καταγγελία γρήγορα και να οδηγήσει τον δράστη, τον αυτούργο σε γρήγορη καταδίκη. Ευχαριστώ κύριε Παπαδοπούλου. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο στόχος της πρότασης μας βρίσκει ομόφωνους. Τελευταία παρακολουθούμε και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες πολλά φαινόμενα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στους κόλπους της ίδιας της Εκκλησίας υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην καθολική εκκλησία τα οποία μας ανατριχιάζουν γιατί εμείς μεγαλώσαμε τουλάχιστον η δική μας γενιά να πιστεύουμε ότι η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία και η κοινωνία πρέπει να σέβονται τα παιδιά και να τα προστατεύουν. Με ανησυχεί σαν μάνα και ίσως προσεχώς σαν γιαγιά σε ποια κοινωνία φαίνουμε τα παιδιά μας. Ιδίω όταν αυτοί οι κόλποι της Εκκλησίας που θα πρέπει να αγκαλιάσουν τα παιδιά είναι οι ίδιοι που βιάζουν τα δικαιώματά τους. Δεύτερο, προχθές διάβαζα ότι σε μια περιοχή στην Τουρκία παιδιά, νεαρές, νεαρά κορίτσια βιάζονται από τους δασκάλους τους σε σχολείο. Και αυτό είναι κάτι που μου προκάλεσε και πάλι τρομερή ανησυχία. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ο διευθυντής του σχολείου ή ο δάσκαλος να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους σεξουαλικά εγκλήματα εναντίον κοριτσιών. Το τρίτο, στην ίδια την οικογένεια υπάρχουν πολλά περιστατικά που ο ίδιος ο πατέρας, στα ελληνικά η λέξη πατέρας, father, εάν αφαιρέσει την πρώτη συλλαβή, το πα, μένει το υπόλοιπο που σημαίνει τέρας. Είναι πολλές περιπτώσεις που ο ίδιος ο πατέρας γίνεται τέρας, δηλαδή ο ίδιος παραβιάζει σεξουαλικά το παιδί του, τη θυγατέρα. Μα ανησυχούν αυτά τα φαινόμενα Νομίζω ότι στι δικέ μα προτάσει ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αγγίξουμε μία πτυχή. Πώς βοηθούμε τον νέο γονιό, τον πατέρα, τη μητέρα, σήμερα, το θεσμό της οικογένειας που δυστυχώς έχει μια πτυχη πω βοηθουμε τον νεο γονιο τον πατερα τη μητερα σημερα το θεσμο της οικογενεια που δυστυχω εχει μια μεγαλη ρευστοτητα και πρέπει να χτίσουμε περισσότερο και σε κοινέ ποινέ και σε πιο αυστηρέ ποινέ, και στην εθνική νομοθεσία και σε στατιστικά δεδομένα και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα διάλογο και με εκκλησιαστικούς παράγοντες και με γονιούς και με δασκάλους για να δούμε πώς μπορούμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βάλουμε το χέρι και να αγγίξουμε στον τύπο των ύλων. Είναι πολλή δουλειά που έχουμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε μόνο σε νομοθεσίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλους δύο ομιλητές έχω στον κατάλογο ομιλητών. Εκτός αν θέλει να προσθεθεί και κάποιος ακόμη, κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών τώρα. Κυρία Μπλινκεβιτσούτε και κύριος Βόσο. Όντως, συμφωνώ και εγώ ότι μια τέτοια οδηγία είναι απαραίτητη και είναι σημαντικό το συντομότερο δυνατόν να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση. Και στη χώρα μου υπάρχουν μεγάλα σκάνδαλα παιδοφιλίας τα οποία αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και γι' αυτό συμφωνώ και εγώ ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να προβλέπει ένα μηχανισμό που θα καταπολεμά την σεξουαλική ε, κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ακόμη και μέσα στην οικογένεια γιατί είναι συχνό το φαινόμενο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης μέσα στον οικογενειακό και το στενό κοινωνικό περίγυρο. Γι' αυτό είναι σημαντικός ένας τέτοιος μηχανισμός. Πρέπει να λάβουμε μέτρα προστασίας ε, του θύματος γιατί το παιδί γίνεται θύμα και κατά τη διάρκεια της ε, ε, διερευνητικής ή ανακριτικής διαδικασίας ενδέχεται το παιδί να υποβάλλεται άλλη μία φορά στο δράμα ε, και να γίνεται νέο θύμα και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Τρίτον, όσον αφορά την παιδική πορνογραφία και τις ιστοσελίδες, εγώ είμαι υπέρ της διαγραφής, της εξάλληψης των ιστοτόπων και όχι μόνο υπέρ της φραγής, διότι η φραγή δεν είναι κάτι το οποίο διαρκεί για πάντοτε. Τέταρτον, η εφαρμογή των διατάξεων είναι σημαντική από τις αρχές ε, επιβολής της τάξης, από τις αστυνομικές αρχές και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ θετικό το ότι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα, διότι μας ενδιαφέρει και να καταπολεμήσουμε την, την ε, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και την διάδοση αυτών των πρακτικών. Και νομίζω ότι μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα του τι επιδιώκουμε να κάνουμε ε, είτε με τη φραγή είτε με την διαγραφή και εξάλληψη των ιστοτόπων ε, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μέτρα προστασίας και για μένα είναι σημαντικό αυτοί οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες ιστοσελίδων να αναλαμβάνουν ε, την ευθύνη για αυτά τα οποία ε, προσφέρουν προς τα έξω και θα πρέπει να φέρουν ε, την ευθύνη. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας ε, στον κόσμο της διαφήμισης και θα πρέπει με ένα τέτοιο κώδικα διοντολογίας να συμμορφωθούν και αυτοί οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Δεύτερον, χρειαζόμαστε διατάξεις που να είναι εφαρμόσιμες και στην πράξη για να μπορέσουμε να διώξουμε αποτελεσματικά αυτά τα αδικήματα. Και είναι σημαντικό να σκεφτούμε αν θα θεωρήσουμε αδίκημα ακόμη και την παρακολούθηση τέτοιων σελίδων στο ε, διαδίκτυο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κλείνουμε κάθε παραθυράκι γιατί σε αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει ε, να ε, επιτρέψουμε ε, την ήπια αντιμετώπιση και θα πρέπει όταν μιλάμε για την επιβολή κυρώσεων να έχουμε ε, ως μέτρα όχι μόνο την, ε, τις τη της ελευθερίας ποινές αλλά και τη δέσμευση περιουσίας ε, και περιουσιακών στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φώστα. Θα κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις λέει η Πρόεδρος πριν ζητήσω από τον κύριο Μολίνο Κόμπο εκ μέρους του Συμβουλίου να λάβει το λόγο. Καταρχήν συμφωνώ με τους συναδέλφους που είπαν ε, ε, ότι η κατάργηση, η εξάλληψη των ιστοσελίδων ε, θα πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Κάτι που δεν μας εξήγησε η Επιτροπή είναι γιατί προτιμά τη φραγή των ιστοτόπων έναντι της εξάλληψης. Εάν το 50% των ιστοτόπων έχουν έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν είναι μια μικρή χώρα χαμένη στο πουθενά είναι ε, ε, ένα σημαντικός εταίρος μας. Γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Όπως επίσης κάτι που είπαν πάλι πολλοί συνάδελφοι, η τεχνολογία δεν είναι η λύση. Δεν πρόκειται η τεχνολογία να προστατεύσει τα παιδιά μας. Τα περισσότερα παιδιά είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης από άτομα του στενού οικογενειακού ή κοινωνικού τους περιβάλλοντος και πολλοί από εμά έχουμε έχουμε γνώση τέτοιων θεμάτων και αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε μέσω της τεχνολογίας. Και βέβαια πρέπει να εξετάσουμε τεχνολογικές λύσεις, αλλά δεν είναι η τεχνολογία αυτή που θα μας προστατεύσει έναντι της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Και τέλος, μια ε, περισσότερο πολιτική παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσημη εκπροσώπηση στο Βατικανό. Δεδομένου ότι ο κύριο Μπαρόζο θα ε, έχει μια ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου με ηγέτε τη Εκκλησία. μου φαίνεται εντυπωσιακό που αρνείται να εκφραστεί επί του θέματο, λέγοντα ότι δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα συζητάμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι σαφώς είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλήσει εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι μια ερώτηση λοιπόν αυτή, είναι ένα αίτημα προς να μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στον κύριο Μπαρόζο. Του τουλεχθέντως θέλω να ζητήσω από τον κύριο Μολίνο Κόμπο να συνεισφέρει και εκείνο με τις παρατηρήσεις του και θα επανέλθουμε στην εισηγήτρια την κυρία Αντζελίλη. Κύριε Μολίνο Κόμπο, έχει το λόγο. Ah, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα σας ευχαριστήσω που με καλέσατε να μιλήσουμε για αυτό την τόσο ενδιαφέρουσα πρόταση οδηγίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιό που παρουσίασε με μεγάλη ταχύτητα, αν θέλετε, την πρότασή της προς το τέλος Μαρτίου. Και έτσι μπορείτε εσείς και το συζητείτε το θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις προηγούμενες Προεδρίες, Σουηδία και την Τσεχία, που μελέτησαν και μία παρεμφερή πρόταση πέρσι, αλλά από τεχνικής πλευράς έχουμε μία βελτιωμένη πρόταση χάρη σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Μιλάμε για φρικτά εγκλήματα. Εγκλήματα κατά του πιο πολύτιμου αγαθού που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο, τα παιδιά μας και τους ανήλικους. Καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί πρέπει να είναι ένα όνο το οποίο πρέπει να σεβόμαστε απολύτως, να μην το εγγίζει κανένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να κατανοήσουμε, μα πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τέτοιου εγκλήματα. Το καλύτερο νέο θα ήταν να μην χρειαζόμαστε μια τέτοια οδηγία. Να λέγαμε όλοι μεταξύ μα, δεν συμβαίνουν τέτοιου είδου πράγματα, τι τη χρειαζόμαστε. Δυστυχώ όμω η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική. Υπάρχουν τέτοιου είδου εγκλήματα, τέτοιου είδου κακουργήματα και πρέπει να πω ότι όλε οι ενέργειες ε, και του Συμβουλίου και των 27 κρατών μελών και τη επιτροπή είναι να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδου εγκλήματα. Του λεχθέντος. Στην πρόταση αυτή προτείνονται πάρα πολλά από νομικής πλευράς ενδιαφέροντα ε, πράγματα από νομικής πλευράς. Όταν μιλούμε για την παιδική πορνογραφία και εικόνες. Αναφέρονται και οι μάγκας, οι ιαπωνικές, τα καρτούν, τα ιαπωνικά, τα κινούμενα σχέδια όπου έχουμε με σαφή ή μη σαφή τρόπο κάποια υπονοούμενα σεξουαλικά. Και τέτοιου ε, είναι θέμα ίσως και πολιτικής αν θέλουμε τέτοιου είδους ε, ε, εικόνες να τις θεωρήσουμε ως πορνογραφικό υλικό. Τώρα, θα πρέπει να μπουν κάποια όρια, κάποια ορόσημα και από ποινική πλευρά τι συμβαίνει όταν ξεπεραστούν αυτά τα όρια. Τι γίνεται όταν ε, έχουμε τέτοιου είδους ε, ερωτηματικά και θα πρέπει για τέτοιου είδους ε, προβλήματα που δημιουργούνται από αυτά τα κινούμενα σχέδια όταν έχουμε παιδιά ή όχι στην εικόνα να το θεωρήσουμε πορνογραφικό υλικό ή όχι. Τώρα, η πρόταση επιτροπής προβλέπει γενικά ποινές, αυτό που προβλέπεται είναι αποδεκτό. Το... Στην πράξη όμως, τι σημαίνει αυτό. Όταν έχουμε ποινικά μέτρα ή αποτρεπτικά μέτρα, το ερώτημα είναι θα ποινικοποιήσουμε μια τέτοια πράξη, θα επιβάλλουμε κυρώσεις 10 ή 12 ε, χρόνια φυλάκιση, διότι με το σύστημα μείωσης των ποινών, ε, τι κάνουμε, το να συζητάμε αν είναι σωστό να φυλακιστεί Κάποιο 10 ε, χρόνια ή 12 χρόνια είναι σαν να συζητάμε αν στην πραγματικότητα θα κρατηθεί ή θα φυλακιστεί 6, 5 ή 3 μήνε. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι εξίσου ενδιαφέρον είναι το θέμα των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκε ε, κάτω από την ε, ηλικία συνένεσης. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις για αυτό το θέμα στην Ευρώπη. Η ηλικία συνένεσης ε, διαφέρει από μία χώρα στην άλλη. Για άλλους είναι τα 18, η ενηλικίωση, για άλλους μπορεί να είναι το 15, 16, το 17. Και τα συστήματα που έχουν ε, ε χαμηλή, μικρή ηλικία συνένεσης είναι αν θέλετε τα πιο δίσκαμπτα. Δηλαδή σε καμία περίπτωση κάτω από αυτή την ε, ηλικία δεν μπορεί να δεχθεί κανείς ε, τέτοιου είδους καταστάσεις. Στην Ισπανία είναι τα 13. Κάτω από τα 13 είμαστε ε, άκαμπτοι. Τι γίνεται με τους άλλους που έχουν υψηλή ηλικία. 15, 16, 17, 18. Εκεί πρέπει κανείς ε, να είναι πιο ευέλικτος διότι ξέρουμε ότι όλο και περισσότερο μειώνεται η ηλικία ε, στην οποία έχουν την πρώτη του σεξουαλική σχέση τα παιδιά. Το 15 ή το 16 είναι κάτι το θεωρητικό αλλά μπορεί ένα κοριτσάκι που δεν είναι καν 15 αλλά 14,5 να έχει σεξουαλικέ σχέσει με το φίλο τη που είναι 16. Και αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί μια φυσιολογική κατάσταση ενώ κανονικά θα πρέπει να ποινικοποιείται. Γι' αυτό λέγω ότι υπάρχει μεγάλη αυξομοίωση της ε, ευελιξίας αναμφίβολα ε, πρέπει να ποινικοποιείται ε, η παιδική πορνογραφία, αυτός ο οποίος έχει τέτοιου είδους πορνογραφικό υλικό πρέπει οπωσδήποτε να ποινικοποιείται διότι με τη συμπεριφορά του υποδαβλίζει αν θέλετε αυτό το εμπόριο το οποίο το εμπόριο της παιδικής πορνογραφίας είναι πραγματικά κάτι το λυπηρό. Και αυτός ο οποίος μπορεί να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους ε, ιστοσελίδες ε, στο ίντερνετ πρέπει να ε, τιμωρείται. Αλλά υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι λέγουν ότι μόνο και μόνο το να έχει κανείς τη διάθεσή του τέτοιου είδους ε, ε, υλικό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υποστεί κυρώσεις. Ο σεξουαλικός ε, τουρισμός επίσης είναι κάτι το οποίο ως πρακτική θέλει να εκριζώσει η Κομισιόν και θα έχει την πλήρη υποστήριξη βεβαίως της Προεδρίας για να προχωρήσει προς αυτή την ε, ε κατεύθυνση. Τώρα, το άρθρο 6 και στα ισπανικά μιλάμε... Και αποπλάνωση, αποπλάνηση ανηλίκων. Ε, δεν μου αρέσει αυτή η μετάφραση, αλλά έτσι λέγεται. Το 10. Επίσης, ε, αναφέρεται στη, στα ασφαλιστικά μέτρα, στα προσωρινά μέτρα και πρέπει να το δούμε το ε, θέμα πιο λεπτομεριακά. Το θέμα επίσης ε, ε, των ε, παραγραφής θα πρέπει να το δούμε. Μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει σε κακοποιηθεί σεξουαλικά μικρό να μπορεί μετά την ε, ενηλικίωσή του να καταγγείλει αυτό το γεγονός και πρέπει να του δίδεται, να του παρέχεται αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, τα χρόνια παραγραφής επίσης πρέπει να το δούμε. Όσον αφορά τώρα την εξωτερική δικαιοδοσία, θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά το θέμα, διότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί η συνεργασία με τις ε, χώρες στις οποίες μία τέτοιου είδους ε, ε, πράξη έχει γίνει. Και κάποιος χ υπηκότητας πηγαίνει στην ψή χώρα ε, κάνει ένα τέτοιο είδους αδίκημα, ποιο είναι το δίκαιο το οποίο θα τον δικάσει. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε και βεβαίως πάντα έχοντας κατά νου το ότι θα πρέπει να μην παίξει κανείς με την υπηκότητά του, με την χώρα διαμονής του για να μπορέσει κάποιος να ξεφύγει. Να ξεφύγει. Θα πρέπει να συνδυαστούν όλα αυτά τα ε, στοιχεία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε πάντα στη λύση η οποία δεν θα είναι η λύση της ατιμορρησίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσουμε, διότι η ατιμορρησία είναι το χειρότερο πράγμα το οποίο μπορεί να συμβεί σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Μέτρα αρρωγής και προστασίας με μεγάλη προσοχή προβλέπονται μέτρα παρέμβασης είναι επίσης κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί και στο ε, Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Το θέμα της φραγής στο ίντερνετ επίσης βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο συζητείται και υπάρχουν αμφιλεγόμενες ε, ε απόψεις. Το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό θα ήταν η διαγραφή τους τι γίνεται όμως όταν προέρχονται τέτοιου είδους ε, ε, σελίδες, τέτοιου είδους περιεχόμενα από χώρε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να μπορέσει κανείς να διαγράψει, να αφαιρέσει από το κομπιούτερ τέτοιου είδους σελίδες θα πρέπει ε, να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της χώρας που στέλνει τέτοιου είδου σελίδε και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για να μπορέσουν ενδεχομένω σε λήψη συμφωνιών να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτά ήθελα να πω σε πρώτη φάση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω τώρα από την εισηγήτρια, που δεν θα είναι και εύκολη, εύκολο το έργο της αυτό, να μας βοηθήσει να κλείσουμε τη συζήτηση. Κυρία Τζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο διότι πραγματικά μπόρεσα να σημειώσω μία προς μία όλες τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι σκόπιμο θα είναι πρώτα-πρώτα να οργανώσουμε μία συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές για να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για το θέμα αυτό και να μπούμε στην ουσία των περισσότερων ε, ζητημάτων που τέθηκαν. Έπειτα, θα ξεκινήσει και η καθ' συζήτηση στην Επιτροπή μας. Ε, δεν περνάω λοιπόν τώρα στο περιεχόμενο της συζήτηση, γιατί δόθηκαν πάρα πολλά στοιχεία, διευκρινήσεις και καλό είναι να τα δούμε με την δέουσα προσοχή και ακρίβεια. Να έχουμε δηλαδή και μια ανταλλαγή απόψεων με τους Σκιώδης. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερω όλου. Ευχαριστούμε κυρία Αντζελίλη, οπότε θα αναλάβετε την πρωτοβουλία να ζητήσετε την συμβολή των σχεδόν εισηγητών. Σας ευχαριστούμε, καλύψαμε και το σημείο 11. Περνάμε λοιπόν τώρα στο σημείο 12 της σημερινής διάταξης. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσια έκθεση που ετησίως μας οδηγεί σε θερμές συζητήσει και ανταλλαγέ απόψεων, όμως το ζήτημα είναι σοβαρότατο, αφορά την καρδιά τη οργάνωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Γκάλ, την εισηγητριά μα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι ότι το ζήτημα δεν είναι απλό. Ούτε είναι και απλό να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση για την έκθεση αυτή. Όπως πέρσι. Πέρσι νομίζω η έκθεση τελικά, όπως προέκυψε από τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις μας, ήταν καλή. Όμως φέτος το όλο ζήτημα γίνεται πιο σημαντικό και πιο ενδιαφέρον. Έχουμε ένα νέο ρυθμό στην πορεία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Δεκέμβριο του 2009 υπάρχει μια δεσμευτική Ευρωπαϊκή Χάρτα, η οποία εκπροσωπεί, θα έλεγα, Μία από τις πιο εκμοντερνισμένε, εξυγχρονισμένε μάλλον κωδικοποιήσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων παγκοσμίω. Φέτο, δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση λοιπόν στο τι έχει συμβεί και τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη, υπό συζήτηση και πώς μπορούμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν ως αποτέλεσμα με αυτό το νέο ρυθμό στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επίτροπος Ρέντινγκ έχει πει πρόσφατα ότι θα μπορούσε να συγκρίνει το επίτευγμα αυτό με το επίτευγμα της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς. Εδώ λοιπόν πραγματικά θα πρέπει να δούμε πώς κατά τον βέλτιστο τρόπο και προς όφελος των πολιτών μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους νέους θεσμικούς, ε, τα νέο θεσμικό πλαίσιο, τις δομές και τους μηχανισμούς που υπάρχουν στη διάθεσή μας πλέον. Υπάρχει λοιπόν η χάρτα αυτή που έχει δεσμευτική αξία. Υπάρχει επίτροπο επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η οποία υπόσχεται συχνή υποβολή έκθεση για, ε, για το σεβασμό, την τήρηση τη χάρτα. και έχουμε και τι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για επιτάχυνση του έργου σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, υπάρχει η πρωτοβουλία των πολιτών που βρίσκεται υπό εξέλιξη, πολύ σημαντικό ο μηχανισμό στον τομέα αυτό, ο οποίο τώρα δημιουργείται και όπω προηγουμένω αναφέρθηκε, έχουμε και την προσχώρηση στη χάρτα που επίκειται. Θα δούμε τι θα σημαίνει αυτό και στην πράξη. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα εργαλεία, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί δίνουν τη δυνατότητα μιας νέας προσέγγισης από τη δική μας την πλευρά. Εγώ διέτρεξα την προηγούμενη έκθεση και μου δημιουργήθηκε το συνέστημα ότι η έκθεση εκείνη ακόμη θα μπορούσε να ισχύει στα συμπεράσματά της. Όμως προτείνω παρόλα αυτά και γι' αυτό ζητώ τη συμβολή σας, τις εμβουλές σας και τη συνεργασία σας και σε αυτό υπολογίζω και στους και εισηγητές. Θα ήθελα να είχαμε μια νέα προσέγγιση εδώ. Τα ζητήματα αυτά να τα εξετάσουμε αυτή τη φορά με, με μια ανανεωμένη ματιά. Μέχρι τώρα η προσέγγιση μας ήταν ιδιαίτερα πρακτική και πραγματιστική. Αλλά επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη όλε αυτέ οι αλλαγέ, επειδή έχουμε όλο αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα ήταν καλύτερο να είχαμε φέτο μια προσέγγιση περισσότερο οριζόντια. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη εντό ολίγου. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα του κατά πόσον οι εκθέσεις μας στον τομέα αυτό θα πρέπει να είναι περισσότερο διορατικές, να βλέπουν προς το μέλλον, τι είδου θέματα θέλουμε να καλύπτουν και πώς. Διότι, εξ όσων γνωρίζουμε, έχουμε την τακτική υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και την Επιτροπή των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε το Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε όλους αυτούς τους υπάρχοντες μηχανισμούς για να ολοκληρώσουμε το τοπίο. Αυτό που σκοπό έχει να ωφελήσει όλου όσους ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α σκεφτούμε λοιπόν τι θέλουμε να περιλαμβάνει μια τέτοια έκθεση και ποιου στόχου θέλουμε να επιδιώκει. Και είναι μια καλή ευκαιρία έκθεση αυτή να διατρέξουμε και του διάφορους μηχανισμούς, να συζητήσουμε τι θα θέλουμε να προκύπτει από αυτού τους οργανισμού και μηχανισμού να συζητήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, των οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Διότι αυτοί θα αναλαμβάνουν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία και τα ερχόμενα χρόνια. Να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, φορέων και των εθνικών καθώς και να συστήσουμε περισσότερο δυναμική δράση και συνεργασία εντονότερη με τις διεθνείς δομές. Βεβαίως, όλα αυτά θα γίνουν σαφέστερα όσο θα πλησιάζουμε και στην προσχώρησή μας στην Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Για τα θεμελιώδη μάλλον δικαιώματα. Όμως πρέπει να σκεφτούμε τι νόημα θα έχουν όλα αυτά για μας και τους πολίτες μας. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε και τα αρμόδια σώματα του ΟΗΕ τα οποία βρίσκονται κοντά μας, χτυπάνε πολλές φορές στην πόρτα μας και τα, τα οποία πρέπει να ενημερώνουμε τακτικά για τις νέες μας αποφάσεις και τους νέους μας μηχανισμούς. Πάντως προσφέρονται πολλές μορφές συνεργασίας μαζί τους. Τώρα, ποιες μορφές συνεργασίας θα θέλουμε να ενισχύσουμε και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και βεβαίως να δούμε και τους φραγμούς, τα εμπόδια που θα θέλαμε να εξελιχθούν. Τι προβλήματα εντοπίζουμε ότι υπάρχουν σήμερα. Τι δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά στη δημιουργία αυτού του τεράστιου τομέα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε εδώ τρία επίπεδα. Από τη μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νομοθετικέ προτάσει, υποβάλλει νομοθετικέ προτάσει προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το σεβασμό τη ε, Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έπειτα τα κρατημέλη και το Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίζουν ότι όταν υλοποιούν κατά την νομοθετική διαδικασία τις προτάσεις είναι συνεπής ως προς την τήρηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έπειτα έχουμε το επίπεδο της υλοποίησης αυτής καθεαυτής. Όταν υλοποιείται ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα, στην εθνική νομοθεσία δηλαδή, όταν μεταφέρεται. Και εκεί πρέπει να υπάρχει συμβατότητα και τήρηση της χάρτας. Πρέπει λοιπόν να δούμε ζητήματα για το πώς μπορούμε να εξετάσουμε και να αξιοποιήσουμε τους μηχανισμούς που προβλέπει πλέον η Λισαβόνα. Πώς θα τους χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ως προς αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα αξιοποιήσουμε την ίδια την Επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα θεμελιώδη μάλλον δικαιώματα. Την ε, χάρτα πώς θα την αξιοποιήσουμε, αλλά και τον οργανισμό. Επίσης θα πρότεινα να προσκαλούμε συστηματικά την Επίτροπο για τα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην δική μας την Επιτροπή για να συζητούμε ζητήματα σχετικά με τον τομέα αυτό. That would be, ε, largely. Αυτά όλα είναι λίγο πολύ όσα είχα υπόψη. Θα ζητούσα λοιπόν τη στενή σας συνεργασία. Και βεβαίω με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η δική σας η οπτική γωνία. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια νέα προσέγγιση προς τα ζητήματα αυτά και να ανανεώσουμε τις συστηματικές εκθέσει που υποβάλλουμε, τις τακτικές εκθέσεις που υποβάλλουμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. have... Ευχαριστώ κυρία Γκάλ. Δύο συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Η κυρία Ντανούκα πρώτα απ' όλα. Yes, thank you, Chair. Το πρόεδρε. Το αναφέρατε ότι χθε κάναμε πολλές συζητήσεις ε, όταν προετοιμάζαμε και προηγούμενες εκθέσεις η Ένα από τα κυρία θέματα ήταν γιατί δεν αναφέρεται στην έκθεση κανένα κράτος μέλος. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν αναφέρουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα για χώρες εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρουμε κάθε χώρα χωριστά. Αλλά όταν συζητούμε για το τι συμβαίνει εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωση αποφεύγουμε να αναφέρουμε το κράτος. Ίσως για να έχουμε πλειοψηφία όταν ψηφίζουμε. Έτσι θα πρέπει να συνεχιστούν τα πράγματα ή θα πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση. Διότι πιστεύω ότι όταν ε, μιλάμε μόνο με γενικότητες και δεν εξειδικεύουμε για καταστρατηγήσεις ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα σε κάποιες χώρες μέλη, δεν, έχουμε, δεν θα έχουμε βελτίωση του όλου συστήματος. Δεύτερη παρατήρηση αναφέρατε τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της υπεύθυνη Επιτρόπου. Θα ήθελα να αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Κάτι που συνέβη πρόσφατα για αυτό το θέμα. Όταν είχαμε με την Επίτροπο Ρέντιν μία ακρόαση, είπε ότι θα υπάρχει ένα μέλος του προσωπικού το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την πολυγλωσία και τα δικαιώματα των μειονοτικών γλωσσών ε, αναφέρθηκε το θέμα αυτό, αναφέρθηκε ο χάρτης, το θέμα το γλωσσικό. Και είπαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να προωθήσουμε τη χρησιμοποίηση των μειονοτικών γλωσσών. Ε, Επίση, πρέπει να πω ότι πρόσφατα ζήτησε συγγνώμη το γραφείο της κυρία Ρέντινγκ διότι χρησιμοποιήθηκε μία μειονοτική γλώσσα. Και υπάρχει συνάδελφος από Λετωνία και ζητήθηκε συγγνώμη γιατί χρησιμοποιήθηκε Ε, στην προετοιμασία και μιας ε, στατιστικής για την ισότητα των φύλων σε μία από τις ιστοσελίδες της Κομισιόν μία, δεν ξέρω, εστονικά ή ρώσικα ίσως και μετά ζήτησε συγγνώμη επίτροπος. Και οι πράσινοι έστειλαν μια επιστολή για αυτό το θέμα, διαμαρτυρώμενοι στην Επίτροπο, αλλά δεν πήραν ακόμη απάντηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα συντονισμού και προσέγγισης και τοποθέτησης της Κομισιόν για τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα. Υποστηρίζω λοιπόν πλήρως την πρότασή της σας να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Έναν ακόμη ομιλητή έχω. Αν θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο, κλείνω τον κατάλογο. Κυρία Μόρβα. Ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να παρακολουθήσω και την έκθεση και να καταλάβω όλο το σύστημα μετά τη Λισαβόνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίω γιατί και εγώ είμαι νομικός και ασχολούμαι με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι ακόμη αρκετά μπερδεμένη όμως για το πώς τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας ε, θα προστατεύονται πιο αποτελεσματικά μετά τη Λισαβόνα. Τι σημαίνει η επικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν του ότι τα κράτη-μέλη μεμονωμένα θα την έχουν επικυρώσει. Τι θα σημαίνει ο χάρτης και οι διάφοροι οργανισμοί που θα έχουν σχέση με τον χάρτη. Και η πρότασή μου προς την εισηγήτρια, ιδίω διότι και οι δύο είμαστε από την Ουγγαρία και η Κίνγκα και εδώ, θα ήταν χρήσιμο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, ένα, γιατί έχουμε ένα παράδειγμα σοβαρής παραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνέβη πρόσφατα. Και θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να εξηγήσει με βάση αυτό το παράδειγμα ποια θα είναι η μεγάλη αλλαγή πριν και μετά τη Λισαβόνα, τι διαφορές υπάρχουν για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το 2006, στις 23 Οκτωβρίου, όπως θα γνωρίζετε, το ΦΙΝΤΕΣ, το κόμμα της εισηγήτριας, ένα κεντρό ουγγρικό κόμμα, οργάνωσε την 15η επέτειο ε, της Επανάστασης του 1956 και ε, ε, στο δρόμο υπήρχαν χιλιάδες διαδηλωτές, η συγγήτρια και εγώ και πολλοί γνωστοί μας και τα παιδιά μας και η αστυνομία ε, επετέθη τους αθώους διαδηλωτές και είχαμε πολλούς ε, τραυματίες, είχαμε προβλήματα και στα μάτια γιατί οι αστυνομικοί προσπαθούσαν ε, χρησιμοποιώντας ακόμη και πλαστικές σφαίρες να μας αποθήσουν πριν από τη Λισαβόνα δεν θα είχε συμβεί τίποτα θα θεωρεί το μια εσωτερική υπόθεση της Ουγγαρίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθήσαμε ε, να επιδιώξουμε διάφορες κατευθύνσεις χωρίς αποτέλεσμα. Και το όλο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θεωρείται ότι έχει καμία δικαιοδοσία και δεν θα μπορούσε να δοθεί καμία απάντηση από αυτού. Θα μπορούσατε σιγά σιγά να κλείνετε την παρέμβαση σας, ρωτάει η Πρόεδρος. Ναι, ξέρω Πρόεδρε ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα που θίγω. Δεν νομίζω όμως ότι μιλώ περισσότερο χρόνο από ότι οι προηγούμενοι ομιλητές. Ελπίζω η ερώτησή μου να είναι σαφής. Κυρία Συγκήτρια, θα μπορούσατε με βάση αυτό το παράδειγμα ποια θα είναι η διαφορά μετά τη Λισαβόνα σε σχέση με το σύστημα που ήσχε πριν από τη Λισαβόνα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μερβάη. Κυρία Φλότχα έχει ζητήσει το λόγο και μετά θα κλείσουμε τον κατάλογο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά μια και η συζήτηση αυτή γίνεται πολύ νωρίτερα σε σχέση με αυτό που είχαμε προβλέψει στη ημερήσια διάταξη, καθυστέρησα λίγο να σα ζητήσω το λόγο. Ζητώ συγγνώμη διότι δεν άκουσα και την παρέμβαση της κυρίας Γκάλ. Από ό,τι κατάλαβα όμως ε, προβλέπει μία δομή που μας απομακρύνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ε, μας απομακρύνει από ένα κατάλογο παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικεντρώνεται σε μηχανισμούς και βελτιώσεις συστάσεων που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε του μηχανισμού μα ε, για την αποτελεσματική εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπω περιγράφονται στο χάρτη και στο, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Υπό αυτή την προσέγγιση λοιπόν μπορώ να πω ότι συμφωνώ απολύτω. Πιστεύω ότι έτσι μπορεί η δική μα συμβολή να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Ταυτόχρονα όμω, διαρωτώ μου κατά πόσο είναι σκόπιμο να εγκρίνουμε κάθε χρόνο μια πολιτική προοπτική η οποία θα είναι σενάρι. Δεν είμαστε Επιτροπή Εμπειρογνωμόντων, δεν είμαστε Εθνική Επιτροπή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, είμαστε Κοινοβούλιο και υπό αυτή την έννοια ε, μία υποτιθέμενη προσέγγιση με βάση παραδείγματο χάρη την αποτελεσματικότητα της πρόσβασης ε, στη δικαιοσύνη των περισσότερων ευάλωτων ατόμων ε, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας θα μπορούσε να αποτελέσει μια επιλογή για φέτος. Μια επιλογή που θα μας επέτρεπε ε, να θίξουμε διάφορα σημαντικά ζητήματα με βάση την ισχυρή μας νομική βάση, δηλαδή την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης σε διάφορους τομείς. Είναι μια προσέγγιση που προτείνεται και από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ετήσια έκθεσή τη και μας επιτρέπει να θίξουμε σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να έχουμε μία διάθρωση που μέσω των οργάνων που έχουν μας και των πολιτικών μας μπορεί να μας επιτρέψει και παράλληλα θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα πιο σκοτεινά σημεία της κατάστασης όταν χρειάζονται κάποιες συστάσεις ή κάποιες ιδιαίτερες προσπάθειες ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει τρόπος να συνδυάσουμε αυτές τις δύο προσεγγίσεις, ούτως ώστε να έχουμε τελικά ένα έγγραφο που θα έχει πολιτική επίπτωση και θα μας δίνουν βάσει αυτού σημασία και το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Αυτός είναι ένας στόχος που πρέπει να επιδιώξουμε. Δεν θα ήταν περιττό, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια συζήτηση σύντομα γύρω από την προσέγγιση αυτή, ούτω ώστε να αρχίσουμε όλοι να εργαζόμαστε με τρόπο στον δυνατόν περισσότερο χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φλότχ και πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί άλλαξε ο χρόνος της συζήτησης του θέματος στην ημερήσια διάταξη. Μάλλον ήταν πολύ γενναιόδωρος ο χρόνος που είχαμε προβλέψει στην ε, ημερήσια διάταξη γιατί να κάνουμε διαλύματα 10 λεπτών ε, κάθε φορά μετά από κάθε θέμα συντομεύσαμε τη συζήτηση. Η κυρία Γκάλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τις διάφορες ε, ιδέες που ακούστηκαν από τους προελίσσαντες. Και θα προσπαθήσω να ανασχολιάσω αυτά τα οποία ελέγχθησαν, γιατί αναφέρονται κράτη-μέλη. Ε, γνωρίζουμε ότι όταν σε μια έκθεση αναφέρονται κράτη-μέλη συγκεκριμένα, δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Σε αυτή την έκθεση έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα. χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα κράτη-μέλη, επομένω να μπαίνουμε σε αντιπαράθεση με άλλους συναδέλφους. Συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει να αναφέρονται τα κράτη-μέλη, αλλά όχι σε αυτή την έκθεση, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν πολλά θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα πρέπει να δούμε ποιος πρέπει να κάνει τι. Να δούμε τι αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι αναμένουμε από τον οργανισμό, ποιο θέλουμε να είναι ο δικό μα ρόλο. Πιστεύω ότι αυτό είναι σημαντικό. να πούμε ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στον Α ή Β τομέα ή στο Α ή Β κράτο μέλο. Τι έκανε η Επιτροπή, τι κάνει η Επιτροπή γενικά. Ο οργανισμό έχει δεδομένα. Γι' αυτό εξάλλου δημιουργήθηκε ο οργανισμός, για να έχει επαρκή αμερόληπτα δεδομένα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Όλα αυτά τα όργανα λοιπόν και οργανισμοί πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε το να κάνουμε μια συζήτηση που δεν θα καταλήγει πουθενά. Γιατί ο ένας από εμάς θα λέει ναι και ο άλλος θα λέει όχι. τέτοιες συζητήσεις ε, που άπτονται θεμάτων ε, και προβλημάτων σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη ε, χρειάζονται πιστεύω σωστά δεδομένα στα οποία να μπορούμε να βασιστούμε. Δημιουργούμε οργανισμούς και όταν λέμε υπάρχει πρόβλημα με ένα κράτο κράτος μέλος, δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον οργανισμό που δημιουργήθηκε ακριβώς για να χρησιμοποιηθεί σε τέτοια περίπτωση, αλλά απλώς λέμε κάτι χωρίς να έχουμε επαρκή δεδομένα αν και, όπως είπα, έχουμε δημιουργήσει τον οργανισμό που θα μπορούσε να μα είχε δώσει τι πληροφορίε βάσει των οποίων θα λέγαμε κάτι. Οπότε τι θέλω να πω, ότι ναι, έχουμε επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε οργανισμούς, έχουμε το συγκεκριμένο οργανισμό. Τι μπορούμε να πούμε τώρα, πώς θέλουμε να λειτουργήσει, τι αναμένουμε. Και αυτό απαντά και στην ερώτηση της κυρίας Μορβάη. Πολλά από τα θέματα που ανέφερε είναι πολύ σημαντικά θέματα. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να δούμε γιατί οι οργανισμοί αυτοί που δημιουργήθηκαν για να κάνουν αυτή τη δουλειά δεν επιτελούν ακριβώς το έργο τους γιατί σε κάποιο σημείο λένε ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος πρέπει να κάνει τι. Χρειαζόμαστε ένα νέο δυναμισμό. Έχουμε ένα δεσμευτικό χάρτη που δεν υπήρχε πριν. Προχωρούμε προς την επικύρωση της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πιστεύω ότι στην έκθεση αυτή πρέπει να πούμε τι προσφέρουμε στους πολίτες με όλα αυτά. Υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες και γι' αυτό θεωρώ σημαντικό Δεν μιλάω ακριβώς στο μικρόφωνο, αλλά ελπίζω ότι με ακούτε καλά. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους οργανισμούς και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να δούμε η νομική βάση που μας προσφέρεται από την Συνθήκη της Λισαβόνας και από τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το χάρτη ε, πώς διαμορφώνουν το σκηνικό για το μέλλον. Αν η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουν πολιτικά μηνύματα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχει σημασία το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Η έκθεση αυτή προβλέπεται για την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Μπορούμε να προσθέσουμε λοιπόν και να συζητάμε όλα τα σημαντικά θέματα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους. Συζήτηση και διάλογος λοιπόν με την Επίτροπο για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα ε, θα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η νέα εκθεσία από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα δημοσιευθεί σύντομα και στις 10 Ιουνίου θα παρουσιαστεί και σε εμά. Στη συνέχεια θα γίνει μια ακρόαση στις 21 και 22 Ιουνίου. και μπορούμε σιγά σιγά να προσθέσουμε νέα δεδομένα. Και γι' αυτό νομίζω ότι η ημερομηνία που έχει προβλεφθεί για την Ολομέλεια τον Νοέμβριο δηλαδή είναι σωστή. Χρειάζομαι τη συνεργασία σας βέβαια γιατί όλα αυτά μαζί θα τα κάνουμε. για να μπορεί το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα με νέο τρόπο μέσα από όλες τις πολιτικές του. και να χρησιμοποιεί όλους αυτούς τους μηχανισμούς προς όφελος των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, uh, σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε και αυτό το θέμα. Τώρα σας προτείνω να διακόψουμε για 45 λεπτά, 40 λεπτά, να επιστρέψουμε στις 11.30 θα κάνουμε κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων για την εμπορία ανθρώπων. Έχουμε μια νέα πρόταση και έχει προβλεφθεί η συζήτηση στις 11.30. Παρακαλώ λοιπόν να έχετε επιστρέψει για τη συζήτηση στις 11.30.

Everybody, I reopen our, uh, our meeting. We have one uh, point of the agenda. Έχουμε ένα ακόμη σημείο στην ημερήσια διάταξη μέχρι το 10.30 πριν το γεύμα. Η εμπορία ανθρώπων κατάργησε της απόφασης πλαίσιο 2002-629. Έχουμε μαζί μας δύο εισηγητές. Το πιο σημαντικό είναι ότι θα έχουμε κοινή συζήτηση βάσει του κανόνα του άρθρου 51 κοινή συζήτηση με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και την δική μας Επιτροπή και οι συζητήσεις αυτές οι κοινές θα λάβουν χώρα εντός των ήδη προβλεπωμένων συνεδριάσεων των δύο Επιτροπών. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η εμπορία των ανθρώπων είναι μια σοβαρή παραβίαση, αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που οδηγεί σε σύγχρονε μορφές βουλεία. Διαβάζουμε συχνά στι εφημερίδες τι πολύ θλιβερέ ιστορίες που πολλές φορές συμβαίνουν στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και να κάνουμε κάτι σχετικά. Και μέχρι τώρα οι πρωτοβουλίε μας δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές. Θα πρέπει λοιπόν ε, να γίνει μια πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου που να καταπολεμά την εμπορία και να προστατεύει τα θύματα. Εν τω μεταξύ θα γνωρίζετε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάστηκε να αναδιατυπώσει την πρότασή της προκειμένου να την ε, αναδιτυπώσει σε πρόταση οδηγία. Έτσι, το Φεβρουάριο του 2010 η Ολομέλεια ενέκρινε ψήφισμα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τώρα θα δούμε σε τι βαθμό οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το ψήφισμα του Φεβρουαρίου έχουν ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη σύνταξη της νέας πρότασης. Συμπροεδρεύω στο σημείο για τη συζήτηση αυτό με την κυρία Σβένσον από την Επιτροπή Γυναικών. Εάν λοιπόν δεν έχει κάτι να προσθέσει, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά πρώτον και μετά στο Συμβούλιο αργότερα. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως αναφέρατε, η Επιτροπή έχει κάνει μια πρόταση στα τέλη Μαρτίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και σαφώς δεν χρειάζεται επεξήγηση, το είπατε και εσείς στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, γιατί το πρόβλημα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει οπωσδήποτε ε, να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά και γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς θέλω να πω ότι είναι απολύτως απαρα... απαράδεκτο να συνεχίσει να υπάρχει τέτοια μορφή δουλεία στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην προηγούμενη θητεία της αλλά και σήμερα θεωρεί την εμπορία ανθρώπων ένα, μία από τις κύριες ε, προτεραιότητές της. Η πρόταση οδηγίας είναι κατά πολύ παρόμοια με την πρόταση για νέα απόφαση πλαίσιο για το ίδιο θέμα που είχε υποβληθεί και είχε συζητηθεί στο Συμβούλιο το 2009. Όπως ίσως γνωρίζετε, η συζήτηση στο Συμβουλίο οδήγησε σε μια συμφωνία επί της αρχής μεταξύ κρατών μελών στο κείμενο, στο Συμβούλιο ΔΕΗ στις 30 Νοεμβρίου πέρυσι. Αυτό το συμφωνημένο κείμενο με κάποιες τροποποιήσεις αποτελεί τη βάση για την πρόταση που υποβάλλεται τώρα. Η πρόταση οδηγίας ε, θα συμπεριλάβει το περιεχόμενο της παλιάς οδηγίας πλαίσιο του 2002 καθώς και το ε, ε, υλικό του σχεδίου συμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, κυρίως ε, τονίζουμε τα σημεία της ενίσχυσης και προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων. Επεκτείνουμε ε, θέματα σε δικήματα που διαπράττονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόβλεψη υψηλότερων και πιο αυστηρών ποινών. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρεται τη 10 Φεβρουαρίου του 2010 για την πρόληψη εμπορίας ανθρώπων. Και με μεγάλη μας ικανοποίηση σημειώνουμε ότι η πρότασή μας είναι πολύ κοντά στις συστάσεις που κάνει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε με την ε, διαπιστωσή μου αυτή. Προς το παρόν δεν θέλω να σας παρουσιάσω λεπτομερώς την πρόταση, απλώς θέλω να πω ότι είμαι πεπισμένο ότι αυτή η πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εκρίζωση και σημαντική μείωση τουλάχιστον του, του εγκλήματος. Θεωρεί η Επιτροπή ιδιαίτερα φιλόδοξη την πρόταση αυτή, διότι ε, έχει ακολουθεί μια προσέγγιση εστιασμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι οι προτινόμενες διατάξεις ε, αποσκοπούν ε, στην υψηλότερη προστασία των θυμάτων και στην πρόληψη αυτών των εγκλημάτων. Ε, προβλέπονται και δυνατότητες ποινική δίωξης μέσω ποινικού δικαίου. δεν μπορούμε μέσω αυτής της οδηγίας να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανάγκης για αυξημένη συνεργασία και εταιρική σχέση με τις χώρες αυτές από τις οποίες συνήθως προέρχονται αυτά τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Θα συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες ε, για την δίωξη, την πρόληψη και την προστασία των θυμάτων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τονίστηκε και στο έγγραφο με τις ε, γενικές κατευθύνσεις που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο πέρυσι το Νοέμβριο. Η πρόταση οδηγίας ήδη έχει υποβληθεί στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει γενικά την υποστήριξή τους για την πρόταση αυτή και το περιεχόμενό της. Κάποιες τροποποιήσεις θα γίνουν, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς να τις δούμε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα ζητηθεί από το Συμβούλιο. Πιστεύω όμως ότι είναι εύλογο να θεωρούμε ότι κάποιες τροποποιήσει που πρότειναν τα κράτη-μέλη θα είναι περιορισμένου εύρους. Στην πρότασή μα, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη συζήτηση σήμερα εδώ, είναι ότι θα είναι μία από τις πρώτες ευκαιρίες ε, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίξει το ρόλο του συνομοθέτη σε τομέα που πριν ήταν τομέα τρίτου πυλώνα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει αυτή τη νέα εξέλιξη και περιμένει με χαρά τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο σε αυτά τα θέματα. Όλα τα θεσμικά όργανα συμφωνούν ότι πρέπει να ενισχύσουμε την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε σχετικά γρήγορα να συμφωνήσουμε για το κείμενο της οδηγίας αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου να λάβει το λόγο. Κύριε Μολύνος, έχετε το λόγο. Eh, eh. Σας ευχαριστώ που μου δείτε το λόγο. Και βεβαίως, όπως και πρώτα σε οδηγίες για την, την προστασία των λύκων από σεξουαλική ε, εκμετάλλευση θα πω ότι ευχαριστούμε την Κομισιό διότι όπως έλεγα και προηγουμένως και σε αυτή την περίπτωση παρουσίασε την πρότασή της πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να πω ότι η Ισπανική Προεδρία ανέκαθεν ζητούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιε πρωτοβουλίε να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατό. Και βεβαίω το έκανε αυτό όχι μόνο επειδή το ζητήσαμε εμεί, αλλά διότι όπω και το προηγούμενο και αυτό της εμπορίας ανθρωπίνων όντων είναι ένα θεμελιώδη σημασία θέμα και δεν ε, μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας την πολιτεία να χάσουμε ούτε ένα λεπτό. Το Νοέμβριο του 2009 υπήρξε συμφωνία του θέματος το Συμβούλιο με κάποιες μικροαλλαγές. Στο δεύτερο άρθρο ε, αναφέρονται των διάφορον ε, τα διάφορα είδη αδικήματος στα πλαίσια αυτού του θέματος. Ακολουθείται η σύμβαση της ε, Βαρσοβίας. Αυτά τα οποία λέγονται επίσης για την ε, εμπορία ζητιάνων ε, ειδικότερα είναι κάτι το ε, σημαντικό διότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται ανθρώπινα άτομα, άτομα για αυτού του είδους το αδίκημα γίνεται λόγος αργότερα ε, χωρίς να είναι περιοριστικός στην ε, περιγραφή των διαφορών ε, ειδών εμπορίας. Όσον αφορά τις κυρώσεις, νομίζω ότι αυτά που λέγονται είναι σωστά. Διορθώνεται ένα τεχνικό σφάλμα το οποίο είχαν αναφέρει πολλές αντιπροσωπείες. Δηλαδή, στο παρελθόν αναφερόταν ότι ανώτατος όριο ποινή ήταν 8 με 10 χρόνια ε, και άλλαξε η διατύπωση, διότι όταν λέμε ανώτατο όριο ποινή 8 με 10 χρόνια, όλοι έβαζαν το 8 και το 10. Δεν είχε καμία ισχύ. Όλα αυτά που αναφέρονται εδώ επίσης μπορούν να ισχύσουν για τους ε, ε, ανηλίκους, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, εδώ επίσης αναφέρεται ένα άλλο θέμα σημαντικό όταν αναφέρονται ασθένειες, η εγκυμοσύνη ξέρετε, δεν είναι ασθένεια η εγκυμοσύνη αλλά ένα, μία έγκυος είναι ένα ιδιαίτερα ευάλωτο άτομο και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης πάρα πολύ σωστά αναφέρεται η ευθύνη και η κυρώσει σύμφωνα με το κάθε νομικό σύστημα. Ξέρετε ότι κάθε νομική έχει διαφορετικό σύστημα. Κάποιοι ε, για το θέμα αυτό ποινικοποιούνται ανάλογα με το αν είναι φυσικά πρόσωπα ή όχι. Επίσης οι ανήλικες μπορούν ε, εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένδικα μέσα, αν δεν το είχαν κάνει όταν ενηλικιωθούν ε, κατά του ατόμου που τους έχει οδηγήσει σε τέτοιου είδους δραστηριότητες και επίσης αναφέρονται τα ένδικα ή εξοδικαστικά μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει κάθε κοινωνία, ε, ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, θέματα στέγασης, ψυχολογικής παρακολούθησης των θυμάτων. Γίνεται επίσης λόγω στα ειδικά θέματα, τα διαδικαστικά ή εξωδιαδικαστικά για την προστασία των ανηλίκων όπως επίσης αναφέρεται και το πολύ σημαντικό θέμα της πρόληψης. Η πρόληψη είναι ένα τυπικό, αν θέλετε, τυπική περίπτωση του, ε, που συμπεριλαμβάνεται στο ποινικό δίκαιο, συμπεριλαμβάνεται εδώ στο άρθρο 15, προγράμματα ενημέρωτης, ε, κατάρτασης των ατόμων που είναι σε επαφή με τα θύματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σωστή η πρόταση εσύ όσον αφορά την πρόληψη. Και τελικά το άρθρο 16 γίνεται λόγος για οργανισμό εποπτείας με απόλυτη ελευθερία στα κράτη μέλη και όπως λέγεται ε, στην παράγραφο 17 ούτως ή άλλως ε, τα κράτη-μέλη έχουν ε, την διαδικριτική ευχέρεια να κάνουν ό,τι κάνουν σύμφωνα με το δικό τους σύστημα, την ομοθεσία του συνήθις, θα αρχίσουμε στα πλαίσια της Προεδρίας να έρθουμε σε επαφή και με το Κοινοβούλιο και όπως ξέρετε η πρόταση αυτή δεν θα ολοκληρωθεί στην ε, διάρκεια της δικής μας προεδρίας, αλλά στην επόμενη στην Βελγική και είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι οι συνάδελφοι της Βελγικής Προεδρίας θα προχωρήσουν το θέμα αυτό, καθώς και το προηγούμενο, με εξαιρετικό τρόπο. Η Βελγική Προεδρία, λοιπόν, θα πρέπει να έρθει και αργότερα σε επαφή με εσά, αλλά και εμεί, όπως είπα, ούτω ή άλλω θέλουμε να κάνουμε τα πρώτα βήματα για να συζητηθεί αυτή η πρόταση. Καλή τύχη σε εσά, καλή τύχη και στην επόμενη Προεδρία και ούτω ή άλλως μπορείτε να υπολογίζετε στην ε, ε, σύνδρομη της δικής μας Προεδρίας και της ε, Ισπανικής Αντιπροσωπείας μετά από την παρέλευση του εξαμήνου. Ευχαριστώ. Τώρα έχουν το λόγο οι εισηγητές η κυρία Λίμπε, πρώτα η κυρία Χατ, η κυρία συγγνώμη Χατ, εκ μέρους των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω να έχει μοιραστεί στους διερμηνείς το κείμενο της παρέμβασή μου, λέει η ομιλήτρια. Δεν το έχουν λάβει οι διερμηνείς δυστυχώ το κείμενο της ομιλήτριας. Ευχαριστώ την Επιτροπή και ιδιαίτερα την Επιτρόπο Μάλμστρομ για την πρόταση που μας υπέβαλε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρετε όλοι ότι η εμπορία ανθρώπων θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα παγκοσμίως και καθημερινά αγωνιζόμαστε για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια είναι μία από τις βασικές αιτίες εμπορίας ανθρώπων και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικά την κατάσταση σε όλες τις πολιτικές, όχι μόνο για το ποινικό δίκαιο, αλλά και για τη μετανάστευση, την κοινωνική πολιτική κλπ. Θα προσπαθήσω με δύο λόγια να εκφράσω τη θέση μου για την πρόταση αυτή. Είναι καλή πρόταση, αλλά λείπουν κάποια στοιχεία στην οδηγία. Άκουσα και του συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και χαίρομαι διότι τονίσαμε το θέμα των παιδιών περισσότερο τώρα από ό,τι στο παρελθόν. Και βέβαια πρέπει να φροντίζουμε την ευημερία των παιδιών και το έχουμε ήδη συζητήσει και στο παρελθόν. Επίσης είναι θετικό ότι ε, υπάρχει νομολογία και υπάρχει δυνατότητα καταδίκης σε ευρωπαϊκά δικαστήρια ε, εγκλημάτων τα οποία διαπράχθησαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης σήμερα φροντίζουμε πολύ περισσότερο τα θύματα και τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Έχουμε υποβάλει μια προφορική τροπολογία για τα θέματα της εμπορίας ανθρώπων Πιστεύω ότι λείπουν κάποια στοιχεία στην πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Παραδείγματος χάρη, όσον αφορά τα εγκλήματα στο διαδίκτυο, διότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να γίνεται με την βοήθεια του διαδικτύου. Χρειάζεται συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και με τους ε, συντονιστές σε επίπεδο κρατών μελών και αυτό το στοιχείο πρέπει να προσθεθεί στην πρόταση. Κάτι άλλο που δεν έγινε αποδεκτό είναι η συγκέντρωση δεδομένων. Ε, υπάρχει πρόβλημα και σε σχέση με την παιδική πορνογραφία. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει σημαντική τεχνογνωσία και θα πρέπει η Europol μαζί με την Frontex και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους. Στο άρθρο, 15 υπάρχει μια πρόταση για εκστρατείες πληροφόρησης στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα οι ενημερωτικές εκστρατείες ε, να διεξάγονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό θα ευαισθητοποιήσει και τα θύματα, αλλά και θα προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε αυτούς που υποβοηθούν σε αυτά τα εγκλήματα. Ξέρουμε ότι συνήθως τα θύματα είναι νεαρά κορίτσια και γυναίκες ε, και τονίζουμε πολύ την ε, πτυχή των παιδιών. Δεν ε, τονίζουμε όμως τις νεαρές γυναίκες και τις γυναίκες όταν μιλάμε για την εμπορία ανθρώπων. Πρέπει να το τονίσουμε για να είναι αποτελεσματική η νομοθετική πράξη. Στην πρόταση προτείνουμε την ποινικοποίηση των δραστηριοτήτων και αυτών που αγοράζουν προϊόντα εμπορίας ανθρώπων. Παραδείγματο χάρη είναι αυτοί που χρησιμοποιούν εργατικά χέρια πάρα πολύ φτηνά ή που ε, χρησιμοποιούν τα προϊόντα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Το άρθρο 15.4 πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι δεσμευτικό, δηλαδή θα πρέπει να θεωρείται ότι ποινικοποιείται και η δραστηριότητα αυτού που επωφελείται από την εμπορία ανθρώπων. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, μιας και είναι παρόντες. Πρώτη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί περιορίζουμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στο άρθρο 9.2. και στο σημείο Γ συγκεκριμένα. Στο 9.1 Γ. Και μια ερώτηση προς το Συμβούλιο. Τι δυνατότητες υπάρχουν να ποινικοποιούνται οι δραστηριότητες αυτών που αγοράζουν τις υπηρεσίες ε, μετά την εμπορία ανθρώπων. Στις 10 Ιουνίου θα γίνει και ένα σεμινάριο για την εμπορία ανθρώπων όπου είστε προσκεκλημένοι. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η κατάθεση τροπολογιών θα έχει προθεσμία όχι στις 2 Ιουνίου, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στις 30 Ιουνίου. Θα σας πούμε όμως πότε θα είναι η ακριβής προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα σας ενημερώσουμε. Θεωρούμε σημαντικό ε, να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό το σεμινάριο και στη συνέχεια να υποβάλουμε τροπολογίες. Θα περιμένω να ακούσω και αυτά που έχει να μας πει η κυρία Μπάουερ και οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε κυρία Χατ. Κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κείμενο αυτό αποτελεί ένα βήμα προόδου και μάλιστα σημαντικό. Συμπεριλαμβάνει έναν τελείως νέο ορισμό, ευρύτερο, που θα τον ε, αξιοποιήσουμε υλοποιώντας την νομοθετική αυτή πράξη. Πολύ χρήσιμο λοιπόν αυτό και για το μέλλον και επίσης καλωσορίζουμε το γεγονός ότι σε σχέση με το προηγούμενο κείμενο το πεδίο των ποινών συμπεριλαμβάνει και την καταναδικαστική επαιτία. Κάτι που ως τώρα δεν έχει οριστεί ως αδίκημα. Είναι μια Δραστηριότητα που έχει δώσει πολύ σοβαρά κέρδη σε όλη την Ευρώπη. Αλλά και σε άλλους τομείς βλέπουμε πολλά σημαντικά βήματα πρόοδου σε αυτή την πρόταση. Επίσης και η θεματοποίηση των παιδιών καλύπτεται από την πρόταση. Και όλα αυτά είναι πράγματα που προσδοκούσαμε από καιρό. Πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μία φορά μόνο θα εξετάζονται στα πλαίσια αυτή τη διαδικασία. και η, βιντεοσκόπηση μια τέτοια συνέντευξη να αξιοποιείται στη συνέχεια της ακρόαση και της διαδικασίας της ποινική. Βεβαίω υπάρχουν ερωτηματικά, υπάρχουν ε, κάποιες αμφιβολίε, κάποιες διατυπώσει θα μπορούσαν να αποσαφινιστούν αλλά αυτά θα καλυφθούν ούτω ή άλλω. Θα ήθελα εγώ από την πλευρά μου να θέσω κάποιες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερωτήσεις που θεωρώ ότι δεν απαντώνται ικανοποιητικά από την πρόταση. Σε ό,τι αφορά την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, καλύπτει την προστασία των θυμάτων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση. Το στοιχείο αυτό λείπει από την πρότασή σας και δεν κατανοώ ακριβώς γιατί. Για ποιο λόγο δεν αναφέρεται κάτι, κάτι που αναφερόταν στην πρόταση 136 μείωση, στη, για το, μείωση του μέγιστου χρόνου ποινή. Ελάχιστη, ελάχιστη ποινή από 6 έως 5 και από 6 σε 5 μάλλον και από 12 σε 10 χρόνια. Αν θεωρούμε ότι αυτή η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι απαράδεκτη, γιατί υπάρχει τέτοια μείωση. Μιλάμε για σοβαρά αδικήματα. Δεν καταλαβαίνω εδώ την μείωση. Τη μείωση από τη μια νομοθετική πράξη στην άλλη. Επίσης υπάρχει και κάτι ακόμη που παραμένει ασαφές. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που το κείμενο αυτό καλύπτει την εμπορία οργάνων. Αλλά δεν είναι απολύτως σαφές τι διαφορετικές διατάξεις θα καλύπτουν το ίδιο θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει εδώ κάποια τροποποίηση για να αποσαφινιστεί. έχω και ένα ακόμη ερώτημα στην πρότασή μας για ψήφισμα. Είπαμε ότι συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει θέση για Ευρωπαίο Επίτροπο για τέτοιο ζήτημα. Υπάρχουν διεθνείς απεσταλμένοι και επιτετραμένοι για τέτοιες περιπτώσεις. Στην Επιτροπή όμως όχι. Εδώ φαίνεται να υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ του έργου των διαφόρων γενικών διευθύνσεων σε αυτόν τον τομέα. Και υπάρχει κάτι ακόμη που θα ήθελα να αναφέρω <clears throat> Αυτό είναι η ηλικία όριο των 18 ετών. Έχω ακούσει πολλά παράπονα από διάφορους εμπειρογνώμονες που λένε ότι η μεθοδολογία αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Λένε ότι είναι παροχημένη, ανάγεται στη δεκαετία του 20 και του 30 και ε, ότι το ηλικιακό αυτό όριο έχει τεθεί από τότε. Εάν λοιπόν εδώ υπάρχει αντίληψη για το τι εννοούμε παιδί ή ανήλικο και πρέπει να έχουμε την ανάλογη συμπεριφορά, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο εντοπισμός ε, του ορίου ηλικίας έχει να κάνει και με τα έγγραφα που στοποιούν την ταυτότητα των παιδιών ή ανηλίκων. Υπάρχουν όμως και μέθοδοι πιο πρακτικές, οι ακτινογραφίες των οστών και των δοντιών για να καθοριστεί η ηλικία. Πολλοί θεωρούν ότι αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ ταπεινωτικές βεβαίως, οπότε πρέπει να ληφθεί και αυτή η πλευρά υπόψη. Ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Έχουμε ακόμα τρεις συναδέλφους που θα ήθελαν να παρέμβουν. Οπότε με τέσσερις ακόμη αγορητές θα κλείσω την, τον κατάλογο αγορητών και μετά τη συζήτησή μας θα ξαναδώσω το λόγο στην Επιτροπή. Πρώτη κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία έχει ως στόχο την προστασία, την ε, καταστολή και την πρόληψη. Θα ήθελα να μιλήσω για την προστασία. Το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε πάντα είναι να βοηθούμε τους ανθρώπους να προστατεύονται και να, επι... να τα... και να βοηθούμε τα θύματα της εμπορίας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε αναφέρεται πολύ λίγο. Αναφέρεται στο ενημερωτικό έγγραφο ότι αυτό δεν είναι μέρος της οδηγίας. Είναι το θέμα της άδειας παραμονής. Η τελευταία οδηγία στην οποία βασίζεται αυτό είναι το θέμα της προσωρινής άδειας διαμονής. Τι σημαίνει αυτό για την προστασία των θυμάτων. Νομίζω ότι υπάρχει ένα κενό σε αυτή την οδηγία. Μπορούμε να βοηθήσουμε με νομική αρρωγή τα άτομα, μπορούμε να βοηθήσουμε με τα άτομα με ψυχολογική βοήθεια, με υλική βοήθεια, με στέγαση, αλλά αν δεν μπορέσουμε να τους εξασφαλίσουμε μια άδεια παραμονής, προσωρινής ή μόνιμης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βοηθήσουμε να τα τα άτομα αυτά να προστατευτούν. Η τελευταία οδηγία μιλάει για την προσωρινή άδεια διαμονή σε συνεργασία με την ε, ε, δίωξη. Και ίσως φοβούνται να κάνουν κάτι τέτοιο τα θύματα. Εδώ συνεχίζεται και λέει ότι υπάρχει δίωξη ακόμη και όταν ε, ένα θύμα δεν θέλει να συνεργαστεί. Άμα βρείτε τον υπεύθυνο έχει καλός, αλλά τι γίνεται σε άλλες περιπτώσεις και τι γίνεται με αυτή την περίπτωση της άδεια παραμονής. Νομίζω ότι εάν το συμπεριλάβουμε αυτό θα βελτιώσουμε την πλωστάσιο της προστασίας και θα επιστρέψουμε στα θύματα να προστατεύονται καλύτερα, διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο ίσως είναι πιο αμφιλεγόμενο, είναι το θέμα της ποινικοποίηση αυτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενώ θύματος εμπορίας. Εάν ποινικοποιήσουμε την πράξη και αυτόν ε, ο οποίος εκμεταλλεύεται μία ιερόδουλη Φερρυπίν, ποινικοποιούμε και την ίδια, το ίδιο το άτομο που παρέχει αυτή την υπηρεσία. Δεδομένου ότι εδώ, εδώ επισέρχονται και άλλα ε, θέματα. Και αν ε, η δουλειά ε, ποινικοποιηθεί, περιθωριοποιείται το άτομο το οποίο είναι και θύμα πολλές φορές. Επίσης, κάτι άλλο που θα ήθελα είναι, είναι όλα αυτά δεσμεστικά ή όχι, δεν το ρώτησε στο Συμβούλιο. Και στην προηγούμενη οδηγία είχαμε ένα ελάχιστο ε, κατόφλι κανόνων που έπρεπε να είναι υποχρεωτική για όλους. Θα ήθελα να μου πείτε τώρα τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση και επίσης με το θέμα της άδειας παραμονής να μου πει η Κομισιόν τι κάνει. Έχουμε και άλλους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο στο μεταξύ. Τώρα η επόμενη μιλήτρια η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ένα θεμελιώδες προκατακτικό ερώτημα σε αυτό το θέμα που συζητάμε είναι πώς βλέπουμε τη διασύνδεση μεταξύ ε, της εμπορίας, ανθρώπ... της εμπορίας ε, γυναικών και παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση και της σεξουαλικής βιομηχανίας και της πορνείας απ' την άλλη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε το να πρέπει να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. από έρευνες ε, και από δικές μου προσωπικές έρευνες ε, με θύματα ε, εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών βλέπουμε ότι οι κύριοι λόγοι για τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και την εμπορία τους είναι η σεξουαλική βιομηχανία και η πορνεία που θεωρούνται κάτι το φυσιολογικό αν θεωρείται φυσιολογικό το να χρησιμοποιούνται οι γυναίκες και να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης οι γυναίκες για σεξουαλικούς σκοπούς στο πλαίσιο της πορνείας και στην ε, βιομηχανία ε, του σεξ, τότε θα υπάρχει συνεχώς ε, ανάγκη για μεγαλύτερη προσφορά γυναικών. Παρότι θεωρείται ότι είναι εργαζόμενες στον τομέα του σεξ, φαίνεται ότι όσο ενδιαφέρον και αν είναι αυτός ο τομέας δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες που να θέλουν να μπουν σε αυτό τον καταπληκτικό κόσμο της πορνείας και θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση και για να ικανοποιηθεί η ζήτηση θα πρέπει να δημιουργηθεί τεχνικά και η προσφορά μέσω της βίας, μέσω της εκμετάλλευσης και μέσω της εμπορίας γυναικών. δεν νομίζω ότι βοηθάμε τα θύματα αν απλώς παράγουμε περισσότερα έγγραφα και κείμενα χωρίς προηγουμένως να εξετάσουμε εις βάθος αυτή τη διασύνδεση. Για την πρόληψη λοιπόν της εμπορίας γυναικών ο καλύτερος τρόπος είναι η πρόληψη της πορνείας και η προστασία των θυμάτων θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αν προσφέρουμε υπηρεσίες όχι μόνο για τον εντοπισμό των θυμάτων και των ε, επιζώντων από την εμπορία ανθρώπων, αλλά κυρίως αν ασχοληθούμε με τις γυναίκες ε, οι οποίες θέλουν να φύγουν από την πορνεία γιατί είναι ένα πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε, ότι οι γυναίκες θέλουν να εγκαταλείψουν τον κόσμο της πορνείας, δεν έχουν υπηρεσίες που να τους ε, παρέχονται. Και αυτό αφορά και την εξαναγκασμένη πορνεία και την κατασυνένεση πορνεία. Δεν λέω ότι η πορνεία θα πρέπει να ποινικοποιηθεί, γιατί θα ήταν σφάλμα αυτό για τις γυναίκες που βρίσκονται στον, στη βιομηχανία της πορνείας. Πρέπει όμως ε, να μάθουμε περισσότερα ε, από τις εμπειρίες άλλων χωρών, όπως η Σουηδία για αυτό το θέμα της ποινικοποίηση των υπηρεσιών πορνείας, και ακόμη και όσοι γνωρίζουν ότι μέσω εντός εισαγωγικών των υπηρεσιών εμπορίας γυναικών αμφισβητούμε το αν ποινικοποιούνται, πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ποινικοποιούνται αυτές ε, οι δραστηριότητε. Επόμενη μιλήτρια, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ Ευχαριστώ τις εισηγήτριες καθώς και τους παρεμβαίνοντες από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό η πρόταση αυτή της Επιτροπής. Είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα στο οποίο θα μπορέσουμε να ασκήσουμε και την δυνατότητα που μας δίνει η συναπόφαση. Και είναι ένα ζήτημα που μας συνερπάζει, νομίζω, εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια. Όλο στο κοινοβούλιο, αλλά και στα εθνικά μας κοινοβούλια. Είναι πολλές οι οργανώσεις που εργάζονται σε αυτό το μέτωπο. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω εδώ την περίπτωση μιας γυναίκας, βουλευτού, η οποία πέθανε πριν από λίγες μέρες, Πάολα Κολόμπος Βέβο, η οποία ήταν συναδελφός μας εδώ πριν από δεκαετία, από το 1996 και ήταν από τις πρωτεργάτριες της Λευκής Βίβλου για κατά της εμπορίας ε, ανθρώπων. Το θυμίζω γιατί ένα αυτό ήταν ένα από τα θέματα που εκείνη πρωτοεσήγαγε ώστε ως θέμα συζήτηση στο κοινοβούλιο μας. Τώρα, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πολύ σωστά θύμισαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι το ζήτημα αυτό είναι σοβαρό, γι' αυτό και εμείς του ζητήσαμε να κάνουν κάποια πρόταση σχετικά. Πολύ σωστά λοιπόν ανταποκρίθηκαν με πρόταση οδηγίας. Κάτι τέτοιο ζητούσαμε και εμείς και κάποιε από τι παρατηρήσει μα όντω ενσωματώθηκαν στη νέα πρόταση. Όμω να θέσω και εγώ κάποιε ερωτήσει. Θα συμμεριστώ κάποιε από τι παρατηρήσει που έγιναν κυρίω για το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα πρόοδου σε αυτό το επίπεδο, διότι πράγματι σήμερα δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα υπάρξει πρόληψη χωρίς ε, ενημέρωση και παρεμβάσει. Υπάρχουν οι εθνικοί φορεί που έχουν τι δυνατότητε παρέμβαση πλέον και μέσω του συντονισμού των δικτύων και των ερευνών. Και θα πρέπει βεβαίως να αντιληφθούμε ως αδίκημα και αυτό που μπορεί να προκύπτει στον κυβερνοχώρο, τον ποινικό όπως έχει ονομαστεί εντός εισαγωγικών. Έχουμε εργαλεία έρευνας και καταπολέμησης και αναζήτησης ανείχνευσης της εμπορίας. Έπειτα, ακόμα και αν έχει εκφραστεί αυτό ως αρχή, θα πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των οικογενειών των θυμάτων της εμπορίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 13. Σε σχέση με αυτό που ζητούσε το ψήφισμά μας, η διάταξη που προβλέπεται στην πρόταση είναι πολύ πιο αδύναμη. Δεν αρκεί εδώ η δράση των κρατών μελών. Τα άτομα αυτά ίσως να πρέπει να στηριχθούν και με την ε, δυνατότητα να έρθουν κοντά τους λόγου χάρη στα θύματα, δηλαδή μέλη της οικογένειάς τους. Δεν υπάρχουν εδώ όμως επίσης καθόλου αναφορές στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Θα πρέπει νομίζω να το θυμηθούμε ότι το ζήτημα της εμπορία το θέτουν πρόταση οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πριν από τα θεσμικά μας όργανα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δυνατότητα αντίδρασης σωστή, εάν δεν έχουμε και μια πρόσκληση προς τα κάτι μελη έκκληση μάλλον, να στηρίξουν τα δίκτυα, τη οργανώσεις που αναλαμβάνουν δράσεις στον τομέα αυτό. Πολλές φορές αυτές οι οργανώσεις είναι που εξασφαλίζουν ε, την προστασία, την ε, κοινωνική ενσωμάτωση, την υποδοχή, την ε, παρακολούθηση των θυμάτων της εμπορίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μια σχετική μνήμα. Και θέλω επίση να καταλάβω και εγώ καλύτερα, όπω είπε η συνάδελφο Μπάουερ, και εδώ παραδέχομαι την άγνοιά μου. Εφόσον δικαιολογείται αυτό ο αποκλεισμό για την ανθρωπιστική παραμονή, κάτι που είναι και αντικείμενο προηγούμενη οδηγία δεν θα πρέπει να εισαχθεί έστω και μέσω ω δικαίωμα. Ή είναι μια έλλειψη τη πρόταση αυτή οδηγία που προσπαθεί παρόλα αυτά να καλύψει ολόκληρο το ζήτημα. Διότι εάν αυτό αληθεύει, εάν δηλαδή πρόκειται εδώ για έλλειψη, για παράληψη, πρόκειται για μια σοβαρή παράληψη και για οπισθοχώρηση. Παναχώρηση μάλλον σε σχέση με τα όσα ως τώρα έχουν αποφασιστεί. Και επίση να πω ότι ο συγητής, μάλλον ο συντονιστή μα. Ε, παρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του της ετήσιας έκθεσης. Είναι σημαντικό για την Επιτροπή να συσχετήσει τη δράση των συντονιστών, των εισηγητών, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, που τα κράτη-μέλη ορίζουν και κάτι που ακόμη δεν είναι ποινικό αδίκημα ίσως, αλλά εγώ θα ήθελα να γίνουν πιο αυστηρε οι ποινέ, έστω οι κυρώσεις και μετά οι χώρες επιμέρου μπορούν να διαλέξουν αν δεν πρόκειται για διοικητικέ ή ποινικέ κυρώσεις, για τα ζητήματα που αναφέρθηκαν και αυτό θα έπρεπε να τονιστεί. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει το λόγο μετά η Επιτροπή. Παρακαλώ λοιπόν να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Η κυρία Αλφάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρίσκω την πρόταση τη Επιτροπή ιδιαίτερα φιλόδοξη. Αλλά θα ήθελα κάποιε διευκρινήσει, ιδίω για το άρθρο 9, στο πρώτο εδάφιο, σε ό,τι αφορά την παράγραφο Β, Γ και Δ. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο για τον οποίο στο άρθρο 9, στο δεύτερο εδάφιο, υπάρχει διάκριση σε σχέση με τα προηγούμενα εδάφια, γάμα και δέλτα του πρώτου εδαφίου, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του αδικήματος. Να δώσω εδώ ένα παράδειγμα για να, καταλα... για να καταλάβετε πού προέκυψε η παρανόηση. Τις τελευταίες ημέρες ακούμε ερωτήσεις για την ε, εκπόρνευση ανηλίκων στην ε, Καμπότζη. Σε αυτούς τους οίκους ανοχής δυστυχώς υπάρχουν ε, συγκεκριμένες μαρτυρίες για κοριτσάκια τριών, τεσσάρων ετών, τα οποία προσφέρονται σε πελάτες που μάλιστα προέρχονται από τις χώρες μας. Εδώ τι δικαιοδοσία θα πρέπει να προβλέψουμε. Δεν θα έπρεπε να είναι αυστηρότατη νομοθεσία για τους καταναλωτές, τους πελάτες αυτούς, οι οποίοι καταστρέφουν τη ζωή των παιδιών. Με ενδιαφέρει λοιπόν πώς η Επιτροπή προβλέπει να καλύψει και αυτό το αδίκημα και πώς θα παρακολουθήσει και την εισαγωγή του αδικήματος αυτού στην νομοθεσία των κατομελών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πουλμπάου Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ συγκεκριμένα θα μιλήσω γιατί πολλές, προτα... πολλές ε, παρεμβάσεις το είπαν. Είναι σημαντική πρόταση, αλλά βλέποντας το περιεχόμενο και άλλων κειμένων στα οποία δουλεύουμε, όπως ε, το θέμα της προστασίας, θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή πώς βλέπουν την εφαρμογή της ε, διαταγής προστασίας των ε, θυμάτων με, αυτό, με αυτή την πρόταση. Διότι πολλές φορές μπορεί να έχουμε θύματα τα οποία έχουν υποστεί τέτοιου είδους παρελόχρηστοι, έχουν υπάρξει θύματα δικτύων εμπορίας, αλλά ξέρουμε ότι τα δίκτυα αυτά εμπορίας είναι ε, διεθνή και ξέρουμε ότι τα άτομα για τα οποία έχει υπάρξει απόφαση καταδικαστική για τέτοιου αδικήματα σε μια χώρα μπορούν να μετακομίσουν και να κάνουν ό,τι θέλουν εκ νέου. Πώς το βλέπεις αυτή την πρωτοβουλία το θέμα αυτό ε, και τι μπορεί να γίνει όταν κάποιος σηκώνεται και φεύγει κάπου αλλού και ξανασυνεχίζει ανενόχλητος. Η κυρία... Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστούμε για την έκθεση αυτή. είναι ένα έγγραφο το οποίο το χρειαζόμαστε. Και η οδηγία αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ερωτήσεις. Κατανοούμε πραγματικά τις αιτίες της εμπορίας των ανθρώπων τον 21ο αιώνα. Η οικονομική κρίση, η μεγάλη φτώχεια, Αυτά είναι προβλήματα που οδηγούν στην εμπορία ανθρώπων. Θα ήταν πολύ σημαντικό ένα από τα μέτρα πρόληψης να είναι και η καταπολέμηση της φτώχειας. Συχνά θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες ή παιδιά όχι μόνο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τρίτες χώρες και αυτές οι γυναίκες ή αυτά τα κορίτσια είναι αντικείμενο εμπορίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεταφέρονται από τη μια χώρα στην άλλη. δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο σταματά μέσα στην επικράτεια μιας χώρας φτάνει πέρα από τα σύνορα και γι' αυτό χρειάζεται αποτελεσματικές τρίτες χώρες. Η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την πρότασή μας όσον αφορά τον συντονιστή. Εγώ συμφωνώ τα άτομα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τέτοιων ατόμων που είναι θύματα εμπορίας θα πρέπει να ε, τιμωρούνται. Θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι και εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δική μας ευθύνη σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Μια τελευταία παρέμβαση από την κυρία Χίρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ω και όδη συγκήτρια από τους φιλελευθέρους χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αυτή τη συζήτηση για αυτή την οδηγία. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και θέματα όπως η επαιτία είναι κάτι το οποίο εμπλουτίζουν την ε, οδηγία αυτή. Η εμπορία ανθρώπων πιστεύω δεν θα πρέπει να θεωρείται μια φυσιολογική διαδικασία και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Στον ίδιο τομέα έχουμε και άλλες δύο οδηγίες, ε, την οδηγία για την σεξουαλική εκμετάλλευση και την παιδική πορνογραφία που συζητήσαμε σήμερα και είναι σημαντικό να δούμε πού βρίσκονται κάποιες κοινέ γραμμές, κάποιοι κοινοί ορισμοί που θα μπορούσαμε ε, να χρησιμοποιήσουμε. Και όπως είπε και η συνάδελφος Σαρτζεντίνη, ε, είναι σημαντικό να δούμε και το θέμα της άδεια παραμονής, γιατί και αυτό συζητιέται στο πλαίσιο του πακέτου για το άσυλο και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ενιαία προσέγγιση σε θέματα τα οποία ε, είναι συναφή. Ε, επίσης, θα ήθελα να αναφέρω κάτι που αναφέρθηκε πολλές φορές, δηλαδή όσον αφορά τους πελάτες των υπηρεσιών που παρέχονται από γυναίκες, γιατί κυρίως οι γυναίκες είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων για το αν θα πρέπει να διώκονται οι πελάτες ή όχι. Νομίζω ότι η ιδέα είναι σωστή. Όταν κάποιος δηλαδή ε, εν γνώση του χρησιμοποιεί υπηρεσίες μιας γυναίκας που είναι θύμα εμπορίας ε, μόνο που θα πρέπει ε, να σκεφτούμε πώς θα γίνεται η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, πώς θα αποδείξουμε ότι ο συγκεκριμένος πελάτης γνώριζε ότι η γυναίκα ήταν θύμα εμπειρίας. Θα πρέπει να ζητάει από την Ιερόδουλο να δείχνει την άδεια παραμονής της, πώς θα ήξερε πραγματικά κάποιος που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ότι ε, μια γυναίκα ήταν θύμα εμπορίας. Καταλαβαίνω τη γενική ιδέα και τη θεωρώ σωστή, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται στην πράξη εφαρμογή αυτής της ε, νομοθεσίας. Γιατί θα πρέπει να έχουμε επαρκή τεκμήρια ε, αν φτάσουμε ε, σε δικαστική διαδικασία για να αποδείξουμε ότι ε, ε, ήταν γνωστό ότι ήταν θύμα εμπορία Μπορεί δηλαδή και η γυναίκα που είναι θύμα εμπορία να φοβηθεί να πάει στην αστυνομία και να καταγγείλει κάτι αν ξέρει ότι θα φτάσει στο δικαστήριο και θα πρέπει να αποδείξει ε, ότι ήταν θύμα εμπορία ενώ δεν διέμενε νομίμως στη χώρα. Ένα άλλο ε, πρόβλημα είναι η εκμετάλλευση ανηλίκων και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι θετικό αυτό το σημείο και εδώ χρειάζεται συνεργασία ακριβώς με αυτές τις ε, τρίτες χώρες να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τεκμήρια στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Χίρς. Ακούσατε πολλές ερωτήσεις. Ε, θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις σας τώρα. Κύριε Πρίμπα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά και σημειώσαμε όλες τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που έγιναν μα έχουν μείνει 7 λεπτά μόνο μέχρι το τέλο τη πρωινή σα συνεδρίασης ε, και δεν νομίζω ότι ε, προλαβαίνω να απαντήσω εκτενώς σε όλε τι ερωτήσει. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση καταρχήν. Η πρόταση αυτή είναι ένα εργαλείο ποινικού δικαίου. ω τέτοιο έχει προετοιμαστεί. Και η πρόταση αυτή όταν θα εγκριθεί δεν πιστεύουμε ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα που έχουν σχέση με την εμπορία ανθρώπων. Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά είναι σαφές ότι ορισμένα ζητήματα, παραδείγματο χάρη αυτά που άπτονται του εργατικού δικαίου, θα πρέπει να ρυθμιστούν από άλλε κοινοτικέ πολιτικέ, πράγμα το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν. Μια δεύτερη γενική παρατήρηση Εδώ έχουμε πάλι μια πρόταση σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα του ποινικού δικαίου μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας και γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη και ορισμένα κράτη-μέλη περισσότερο από ό,τι άλλα κράτη-μέλη διστάζουν πάρα πολύ στο να αφήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει ρυθμιστικές διατάξεις σε αυτό το τομέα του ποινικού δικαίου. Είναι μια οδηγία την οποία προτείνουμε και πολλά θέματα θα πρέπει να αφαιθούν στα κράτη-μέλη για να αποφασιστούν ως προς τις λεπτομέρειές τους. Ε, του λεχθέντος, συμφωνούμε με τα περισσότερα από όσα αναφέρθηκαν από τα μέλη των επιτροπών σας. Αναφέρεται και το θέμα του διαδικτύου και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό αντικείμενο μιας οδηγίας που ασχολείται με την εμπορία ανθρώπων και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα για το πώς θα καταπολεμήσουμε δηλαδή τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Πολλά από τα σημεία που συζητήθηκαν τώρα συζητήθηκαν και στο προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε την σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η ανταλλαγή δεδομένων και θέλουμε να βελτιώσουμε τα δεδομένα και γι' αυτό είμαστε σε επαφή με τη Eurostat για να έχουμε καλύτερα στατιστικά δεδομένα. Αλλά αν δεν έχουμε επαρκή δεδομένα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε μια προσπάθεια νομικής ρύθμισης του προβλήματος. Ε, επίσης, ε, οι εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι κάτι που είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει επιπροσθέτως, εκτός δηλαδή από, την, από τα νομοθετικά μέτρα που θα προτείνουμε. Για την ερμηνεία συγκεκριμένων άρθρων έγιναν αρκετέ ερωτήσει, ε, γιατί αφήσαμε περισσότερο χώρο στα κράτη-μέλη. Τα έχω σημειώσει, αλλά δεν θα σα απαντήσω λεπτομερώ σήμερα για όλα αυτά. Παραδείγματο χάρη στο άρθρο 9 παράγραφο 2 και στο άρθρο 15 παράγραφο 4 θεωρούμε ότι η πρότασή μας αντικατοπτρίζει το εφικτό Σε πολλά σημεία της πρότασης θα θέλαμε να προχωρήσουμε περισσότερο, αλλά δεν έχει νόημα να υποβάλουμε μία πρόταση ε, όπου θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα ε, μεγάλη αντίσταση από τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό έχουμε καταλήξει σε κάποιες διατάξεις που αφήνουν κάποιο πεδίο ελεύθερο στα κράτη-μέλη. Ένα άλλο ερώτημα τώρα για ε, τις μέγιστες ποινές ε, που έχουν ε, περάσει από 10 στα 12 χρόνια. Αυτό αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές καταστάσεις που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Σε ορισμένα κράτη-μέλη η ποινή 12 ετών θεωρείται τόσο υπερβολικά υψηλή που ακόμη και για αυτού του είδους τα εγκλήματα που κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι σοβαρό έγκλημα δεν θεωρείται αποδεκτή σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Ένα άλλο θέμα το οποίο πολλοί βουλευτές ε, έθεσαν και είναι εύλογο σημείο. Αυτά που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής, με θέματα ασύλου ε, και παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχουν θέματα που θεωρούμε ότι καλύπτονται από νομοθεσία σε διαφορετικά πεδία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναβάλουμε εμείς τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Μία από τις οδηγίες ε, στα θέματα εργατικού δικαίου μπορεί να αποτελέσει ένα από τα βήματα για να προετοιμαστεί σχετική νομοθεσία σε αυτούς τους τομείς. Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διορισμού συντονιστού σε υψηλό επίπεδο για θέματα εμπορίας ανθρώπων και η διαδικασία πρόσληψης ενός ε, συντονιστού θα χρειαστεί κάποιους μήνες. Έχει ξεκινήσει όμως αυτή η διαδικασία και θέλουμε να εντείνουμε τις εργασίες μας σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα και να συντονιστούμε καλύτερα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο διεθνές επίπεδο. Ελπίζω ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα μήνυμα για το πόσο σοβαρά παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως συμφωνούμε με τις απόψεις ε, που αναφέρθηκαν ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν και στο άρθρο 15 παράγραφο 2 νομίζω ότι το αναφέρουμε αυτό. Και ξέρουμε ότι η νομοθεσία είναι ένα πράγμα, η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι ένα άλλο πράγμα. Και δεν έχουμε ψευδεστήσεις επ' αυτού. Δεν θα είναι πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήγει σε μια νομοθεσία και μετά δεν γίνεται τίποτα στην πράξη. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας αφού εγκριθεί αυτή η οδηγία και αυτό δεν σημαίνει μόνο μεταφορά της οδηγίας σε εθνικό δίκαιο αλλά και αποτελεσματική εφαρμογή της. Αλλά ακριβώς αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να υπερβάλλουμε στο στάδιο αυτό διότι δεν έχουμε την αποδοχή των κρατών μελών και των κυβερνήσεων και της κοινή γνώμης γενικότερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί σίγουρα να προσφέρει ε, ε, τα πάντα σε αυτόν τον τομέα. Τελικά κάποιες εθνικές αρχές ε, θα πρέπει να αναλάβουν την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι διερμηνείς πρέπει να διακόψουν. Λυπούμε. Αλλά ούτως ή, βάλω, άλλως τα θέματα τα οποία δεν απαντήθηκαν θα απαντηθούν. Αν επιθυμείτε μπορείτε να αποστείλετε γραπτό απαντήσεις σας και οι εισηγητές μπορούν επίσης να απαντήσουν. Παρακαλούμε τους διερμηνείς να μείνουν ακόμη τρία λεπτά, ώστε κάθε εισηγήτρια να μιλήσει ακόμη για ένα μισή λεπτό. Η κυρία Χατ, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα απλώ να πω το εξή. Κύριε Σαρτόρη, μίλησε για ποινικοποίηση των πελατών. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο εδώ με πορνεία. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάποιος υποψήφιος για να θεωρηθεί ύποπτος αδικήματος όχι μόνο όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μιας πόρνης αλλά εάν εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε θύμα εμπορίας. Νομίζω ότι αυτά όλα τα θέματα καθώς και την ε, παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών θα πρέπει να τα ξαναδούμε και έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα τρομερό πρόβλημα και μία μία πραγματική μάστιγα για το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα να το ξαναεξετάσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάουερ, νομίζω ότι έχουμε και χρόνο και άλλες δυνατότητες να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα αυτό και περιμένω την επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε για να παρέμβω. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρία και θα συνεχίσουμε σήμερα το απόγευμα στις 3. Ευχαριστώ συνάδελφοι, καλή όρεξη.